Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι 9 και 6. Θέλουμε αρκετό χρόνο για την ακρόασή μας και για όλες τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, οπότε να ξεκινήσουμε αμέσως. Ε, έχουμε την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας Τετάρτη πρωί, Τετάρτη απόγευμα και Πέμπτη πρωί. Και να ξεκινήσω. Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την ανάληψη καθηκόντων από τη Νέα Επιτροπή. Είναι πανέτοιμη να αναλάβει δράση. Δεύτερο σημείο, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ένα πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2030. Πολύ σημαντικές αποφάσεις σε πολύ σημαντικούς καιρούς. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται στους φακέλους σας. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορεί να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω αλλαγές. Δεν βλέπω να έχετε παρατηρήσεις. Προφανώς γιατί ό,τι άλλο θέλετε να προσθέσετε στα διάφορα την Πέμπτη. του Προέδρου. Να πω πολύ Κοπ COP20 και συνεισφορά της ΙΤΡΑ είναι πολύ σημαντικό συνάδελφοι. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των συντονιστών, μια ανάλογη ομάδα ε, μελών της ΗΤΡΕ, με εισηγητή της ΙΤΡΑ και τους σκιώδης ε, ετοιμάσαμε ένα κείμενο συμβιβαστικών λύσεων το οποίο θα ε, μοιραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση. Βρίσκεται στους φακέλους Βάσει της διαδικασίας των περασμένων ετών, η συνεισφορά της ΙΤΡΕ θα πρέπει να αποσταλεί και στον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΝΒΗ, η οποία Επιτροπή θα ψηφίσει σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα, συνάδελφοι, και θέλουμε να έχουν και τη δική μας την τοποθέτηση. και προφανώ να ληφθεί υπόψη να καταγραφεί. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, υποθέτω ότι μπορώ να αποστείλω τη συνεισφορά μα στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Να αποστείλουμε την δική μας μοδότηση λοιπόν στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Να ξεκινήσουμε, να περάσω απευθεία στο σημείο 3. Δημόσια κρόαση με θέματα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τη υπό συνθήκες Εσωτερική ενεργειακής αγοράς βάση της μελλοντική ενεργειακής αγοράς που θέλουμε να διαμορφώσουμε βέβαια, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία της και τα κράτη-μέλη, οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων, πρόεδροι και πρωθυπουργοί, υπεσχέθησαν το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι το τέλος του 2014 να υπάρχει αυτή η εσωτερική αγορά. Εξ όσων εγώ μπορώ να δω, έχουμε δύο μήνες για να την ολοκληρώσουμε την αγορά αυτή. Τέλος πάντων, να σοβαρευτώ. Και είναι σοβαρό το θέμα. Η εσωτερική ενεργειακή αγορά σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Τι χρειαζόμαστε ακόμα. Είναι προφανές υποδομές, οι οποίες δεν έχουν περατωθεί, διασυνοριακές διασυνδέσεις, τις ανάλογες αποφάσεις για την εμπορία ενέργειας και την, αποστο... την τροφοδοσία σε ενέργεια ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με Κωδικού λόγω χάρη για την ενέργεια ή προγράμματα στήριξη για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας που να μπορούν να είναι συγκρίσιμα εάν θέλουμε τέτοια εμπορία ενέργειας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σταδιακά να καταργήσουμε τη ρύθμιση των τιμών στα κράτη-μέλη. Ιδάλλως, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε απελευθερωμένο εμπόριο στις αγορές μας. Δεν είναι απλό, το γνωρίζουμε. Τα κράτη-μέλη μας δεν μπορούν εύκολα να λάβουν μια τέτοια απόφαση, αλλά έχουμε και τον τριμερή διάλογο για την ενέργεια, μιλάμε για την ασφάλεια της ε, προσιτές τιμές, την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Να πω το εξής, ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι παρόλα αυτά η ασφάλεια. Χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αλλά δεν θέλω να υπονομεύσω τα δύο στοιχεία που είναι εξίσου σημαντικά. Σε αυτή τη φάση όμως θα μιλήσουμε για τη στρατηγική μας, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την έκθεση που ετοιμάζει ο κύριος Σαουντάργας ως εισηγητής. Ε, και με τη συμμετοχή βεβαίω των σκιωδών εισηγητών. Είναι η πρώτη μα ε, συμμετοχή στην όλη συζήτηση, στη φάση αυτή, ε, για την ενεργειακή ασφάλεια. Η ενεργειακή ασφάλεια θα είναι πάντοτε μία από τις μείζονε αρμοδιότητες και δραστηριότητε της Επιτροπής μας. Είναι η πρώτη μας, μάλιστα, έκθεση στη νέα θητεία της Επιτροπής Ήτρε πολύ σημαντική για την Ευρώπη, για όλα τα κράτη και βεβαίως και υπό το φως της κρίσης στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Ο Ζακ Ντελόρ και εγώ όταν προτείναμε στο σώμα αυτό πριν από τέσσερα χρόνια την ενεργειακή κοινότητα, εδώ στο Κοινοβούλιο λοιπόν, ε, που στήριξαν οι συγητές και οι σκιώδεις εδώ, με την κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, τον, την κυρία Σαβέλα και άλλους. Με τη συμμετοχή λοιπόν όλων αυτών η πρόταση αυτή είχε γίνει αποδεκτή. Τώρα προς το τέλος έχουμε τουλάχιστον μία συνέχεια, μία διάρκεια στο χρόνο αυτής της ενεργειακής κοινότητας και την εξέλιξη της σε ενεργειακή ένωση. Η ίδια ιδέα υποκρύπτεται εδώ με κάπως διαφορετικό σλόγγαν, ε, σύνθημα δηλαδή, λίγο διαφοροποιημένο, διότι είναι πιο εντονή έκφραση η Ενεργειακή Ένωση. Αλλά εδώ έχουμε και ειδικό ε, πρόεδρο στην Επιτροπή μας για τα θέματα της Ενεργειακής Ένωσης. Οπότε αυτή μας είναι η πρώτη ε, προσέγγιση του όλου θέματος. Για τους σκοπούς της Ενεργειακής Ένωσης, το πλέον σημαντικό θέμα θα είναι προφανώς η ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της συνεδρίασής μας, είναι μεγάλη μας χαρά να μπορούμε να υποδεχτούμε ε, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, καλώς ήρθατε και καλώς ήρθατε και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την δημόσια ακρόαση, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και στον ιστοτόπο του Ευρωκοινοβουλίου, στο διαδικτύο. Μετά δίδεται ζωντανά. Να ζητήσω από τον εισηγητή μας, θέλετε να τοποθετηθείτε στην αρχή αυτής της ακρόασης. Εσείς αποφασίζετε. Θέλετε να κάνετε κάποια εισαγωγικά σχόλια. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που παρουσιάσατε τόσο σαφώς ε, την κατάσταση. Θα ήθελα απλά να καλωσορίσω τους διακεκριμένους ομιλητές. Ε, περιμένω να ακούσουμε προσοχή τα όσα θα πούν. Ήδη κύριε Πρόεδρε αναφέρατε τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν. Μία σύντομη παρατήρηση τι πρέπει να γίνει η ενεργειακή ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα μία στρατηγική. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ένας βασικός σοβαρός πυλώνας της Ενεργειακής Ένωσης όπως αναφέρατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και αναμένω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Σημαντικό το ότι βεβαίως μετά θα συνοψίσουμε και θα κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, να παρουσιάσω τους ομιλητές να σας ενημερώσω πως έχουμε 3 ώρες και ένα τέταρτο στη διάθεσή μας 12.30 πρέπει να τελειώσουμε χωρίς διάλειμμα δύσκολο για εμένα αλλά θα προσπαθήσω αλλά για κάθε ομιλητή θα ήθελα να σας παρακαλέσω αγαπητοί φίλοι από όλη την Ευρώπη έχετε 10 λεπτά για μια αρχική τοποθέτηση, μετά 20 λεπτά για ερωτήσεις ε, και απαντήσεις. Και αν είστε πάρα πολύ, ε, ίσως λίγο παραπάνω και μετά θα απαντήσετε και τις ε, ερωτήσεις. Και εξαρτάται ε, βεβαίως και από τον αριθμό των ερωτήσεων. Αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Ρώμας Σβέντας είναι ο πρώτος από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Βίλνιους ε, στην Λιθουανία. Και η παρουσίαση είναι οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, μαθήματα και νέες προκλήσεις. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι για μένα μια τιμή που έχω την ευκαιρία να μιλήσω στο εκλεκτό αυτό ακροατήριο σήμερα πιέζει ο χρόνος. Αλλά ξέρετε, ε, ε, έχω προσπαθήσει ε, επί μια εικοσαετία να υπηρετήσω την οικονομική διπλωματία. Τώρα όμως είμαι ανεξάρτητος, ε, είμαι πανεπιστημιακός εδώ και τρία χρόνια. Ξέρω επομένω τι σημαίνει πίεση χρόνου και οπότε και θέλω να σας επισημάνω τρία τεινά. Η υπηρεσία διεθνή ατομικής ενέργειας θεωρεί ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι η αδιάκοπη διαθεσιμότητα των ε, ενεργειακών πόρων σε κάποια εύλογη τιμή και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει ποικιλία στην ε, παροχή αυτής της ενέργειας οπότε έτσι να υπάρχει πρόσφορα όμως δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα το να έχουμε μία εξωτερική σχέση αν ε, ο προμηθευτής και ε, ο καταναλωτής έχουν σχέσεις που διέπονται από διαφάνεια τα προβλήματα ξεκινούν όταν ε, αυτός ο οποίος έχει τους πόρους δεν διακρίνεται από τις δημοκρατικές του αρχές και καταχράται τις ε, δεσπόζουσες θέσεις τη για σκοπούς ε, πολιτικής. Οπότε επίσης έχει κάποιους στόχους πολιτικούς, γεωπολιτικούς, οπότε τότε δεν αποδίδει δεν η οικονομική λογική. Η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας αποδεικνύει το ότι η πολιτική κατησχύει της οικονομίας. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό μπορεί να το διαπιστώσουμε από πολλά στοιχεία όπως το ότι κόβουν την παραχή ενέργειας, δεν έχουν τιμολογιακή πολιτική διάφανη, ε, έχουν διάφορα προγράμματα ενδιάμεσα όσον αφορά την παροχή του φυσικού αερίου, οπότε έχουμε τότε εξάρτηση και ε, ε, έχουμε επίσης την ε, άσκηση επιρροής από πλευράς ε, Μόσχας σε πολλές σημαντικές χώρες. Άρα για ποιο λόγο το γίνεται αυτό για να κυριαρχήσει, για να κυριαρχήσει στις χώρες που ανήκαν κάποτε στο Σοβιετικό μπλοκ για να γίνει παγκόσμια δύναμη. Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημοκρατικό σύστημα και την οικονομία της αγοράς. Αυτό που θέλει το Κρεμλίνο να καταργήσει τη δημοκρατία και τον φιλελευθερισμό, ε, η Ρωσική Ομοσπονδία ε, δεν διακρίνεται από ένα πολιτικό σύστημα δημοκρατικό, καταχράται ακριβώς ε, των ενεργειακών πόρων που έχει και επομένω χρησιμοποιεί την ενέργεια για στόχου πολιτικού. Το πρώτο μήνυμα επομένω είναι ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θέλει να αναστρέψει ε, τον δημοκρατικό μετασχηματισμό και θα θέλει κάποιε χώρε να του οδηγήσει σε κάποια φαιά ζώνη όπου να έχουμε έναν αναποτελεσματικό ε, πλουραλισμό και πολιτική που να καθορίζεται από την κυρίαρχη δύναμη και ε, σας παραπέμπω στο, στο, όσα έχει γράψει ο Σάμιουλ ε, Χάντικτον και ο Τόμας Κάροδερς. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι θα πρέπει τώρα να σας ε, ε, παραπέμψω στον χάρτη που αποτυπώνει την ρωσική δύναμη Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Βαλτικέ χώρε. Όλε αυτέ οι χώρε διέπονται από κάποιον κοινό παρανομαστή. Το ότι δηλαδή είναι όμορε τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο επόμενο χάρτη τώρα που μπορείτε να δείτε σας δείχνει πώς εφαρμόζει την πολιτική, οικονομική και στρατηγική ισχύ η Ρωσία. Και άλλος χάρτης, ο οποίος ε, σας δείχνει το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι ισχύς της πληροφορίας και της διπλωματίας. Οπότε έχουμε τώρα ε, μια κατάσταση πολέμου του ορμαζομένου υβριδικού πολέμου. Η ενέργεια ε, είναι ένα από τα μία από τις πτυχές αυτού του βρυδικού πολέμου και χρησιμοποιείται όχι μόνο σαν ένα εργαλείο, σαν ένα μέσο άσκησης πολιτικής, αλλά επίσης και σαν όπλο. Με το Nord Stream και το South Stream αφημικίνους αγωγούς προσπαθεί να ε, εξασφαλίσει το εισόδημα από τη Δύση η Ρωσία και επίση να κατησχίσει των χωρών κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε επομένω αυτού του δύο ενεργειακού ε, πυρηνικού σταθμού σε Λευκορωσία, στο ήταν λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από το, τα σύνορα με την Λιθουανία. Και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο αποτελεί μια πάρα πολύ ακριβή προσπάθεια, ούτω ώστε να ε, να αντιθασέψουν τις ε, χώρες της Βαλτικής. Επίσης έχουν τα, τα δικά τους έργα, τα δικά τους project, δηλαδή θέλουν να έχουν ε, εναλλακτική ε, παροχή ενέργειας σε κεντρική και ε, Ανατολική Ευρώπη. Αυτό θα το σταματήσει η Ρωσία. Και οπότε το δεύτερο μήνυμα είναι ότι ακριβώς κάθε τέτοιο έργο ή πρόγραμμα που αφορά την ενέργεια έχει σταδιακή σημασία και προσπαθούν με κάποιο είδους επίθεση πληροφορίας να το αμαυρώσουν ούτως ώστε να το καταστρέψουν πολιτικά. Και έχουμε επομένω τέσσερις τέτοιες ε, κατευθύνσεις που παίρνουν, δηλαδή συγκρούσεις με την τοπική κοινωνία, ε, ε, να καταρρεύσει η πριβολική αξιολόγηση, η ασφάλεια και η οικονομική ωφέλεια του έργου και για το συστολιθικό αέριο. Επίσης έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και έχουμε επίσης ε, κακοδιαχείριση. Επίσης, αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν είναι ε, οι νέες πυρηνικές δυνάμεις της ε, περιφέρειας να, να παγώσουν. Και αυτό θεωρήθηκε σαν μια επίθεση σε, σε ένα πρόγραμμα θεμητό κατά τα άλλα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το κάνανε από τότε που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και θα το συνεχίσουν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα είδου διαφάνεια και αυτό αφορά ε, το από πού βρίσκουν τα χρήματα για τέτοιου είδους εκστρατείε τις οποίες ε, διεξάγουν. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κρατημέλη θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και θα πρέπει να λάβουν μέτρα ε, προληπτικού χαρακτήρα. Κυρίε και κύριοι, η ανακοίνωση επιτροπή όσον αφορά την ε, ενεργειακή ασφάλεια ε, έρχεται πάνω στην ώρα και επίσης είναι πάρα πολύ ε, σφαιρική και καλύπτει πολλές προτινόμενες δράσεις οπότε θα πρέπει να σας αναφέρω το θέμα του πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προσφορά φυσικού αερίου και του ρομπινού αερίου και σας λέω ότι αισθανόμαστε περήφανοι γιατί είχαμε τον πρώτο τερματικό σταθμό ε, στην στην Πέντα, το λιμάνι της Λιθουανίας και οπότε εδώ πέρα έχουμε ε, 4 BCM φυσικού αερίου ετησίως. Και ξέρετε πώς ονομάζεται αυτός ο τερματικός. Έχει το όνομα Ανεξαρτησία. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, το το μήνυμα είναι το εξή ότι η βασική πρόκληση της στρατηγικής για την ασφάλεια ε, δεν θα το αναζητήσουμε, θα το βρούμε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κλειδί είναι το υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά κρατών μελών. Θα πρέπει να αναλάβουν δράση τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να ε, τα καταφέρουν και ε, κατά τα άλλα πρόκειται για άσκηση επιχάρτου. το South Stream την Gazprom είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να παρακάμψει τον Ευρωπαϊκό Ναμπούκο το 10 Σεπτέμβριο, ένα κράτος μέλος, δήθεν χωρίς να το περιμένει κανείς, ε, σταμάτησε την ε, παροχή φυσικού αερίου για την Ουκρανία. Η χώρα μου ε, έχασε έναν πάρα πολύ στρατηγικό επενδυτή όσον αφορά το σχιστολιθικό αέριο και σταμάτησε το, το όραμα της ε, πυρηνικής ενεργείας. Γιατί ε, δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Οπότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αγορά μέχρι το 2014, είχαμε πει, αλλά αυτό δεν το καταφέρουμε. Ώστε να υπάρχει εσωτερική ισχυρή ενεργειακή αγορά, θα είμαστε αδύναμοι και γι' αυτό απευθύνουμε σε εσά. Και παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε την ε, επιρροή σας, να καταβάλλετε πάσα προσπάθεια για να εξασφαλίσετε το ότι δεν θα μείνει στα χαρτιά η στρατηγική για ενεργειακή ασφάλεια. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερη δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι αυστηρότερο όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία. Κυρίε και κύριοι, σε αυτή την εισήγηση σα ετώνησα τι τρει προκλήσει σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Πρώτον, χρησιμοποιείται η ενέργεια για την καταπίεση ει βάρο δημοκρατία και φιλελευθερισμού. Δεύτερον, το ότι ο ενεργικός τομέας υφίσταται συνεχώς σε πληροφοριακές ε, ε, ε, επιθέσεις από εκστρατείες ενημέρωσης και την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Όλα αυτά μας δείχνουν στο ότι δεν είναι θέματα μόνο ε, Κατασκευή, είναι θέμα τεχνοκρατικό, είναι θέμα της αγοράς και της οικονομίας, είναι θέμα διεθνών σχέσεων και πολιτική. Άρα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί μια κατηγορηματική ε, απάντηση. Η απάντηση ε, βρίσκεται στην έννοια της αγοράς, της, συγγνώμη, της Ενεργειακής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, σχετικά με αυτό δεν θα πρέπει να βάζουμε ερωτηματικά, δεν πρέπει να ρωτάμε το αν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να ρωτάμε ακριβώ τι θα γίνει και πότε θα γίνει. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστούμε για τις ιδέες αυτές που μας δώσατε, για την ενέργεια ως πολιτικό όπλο, όπλο πολιτικής, για τους ε, κανόνες της εσωτερικής αγοράς και τις διασυνδέσεις που είναι πολύ σημαντικές, ε, σημαντικοί μάλλον, και για τις ε, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πρέπει να παραμείνουν ε, λόγια στο χαρτί, αλλά να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα. Η Ενεργειακή Ένωση είναι μια απάντηση. Σας ευχαριστώ και πάλι και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ευθύς αμέσως. Κύριε Σαουντάργκας, θέλετε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε για αυτή την ε, σφαιρική παρουσίαση των απειλών που έρχονται από Ανατολές. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Στο τέλος της παρουσίασής σας είπατε ο και δώσατε έμφαση στο ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Βούληση να λάβει μια νέα κατεύθυνση προς την Ενεργειακή Ένωση. Ήθελα να ρωτήσω η ενεργειακή στρατηγική και οι σχετικές μας προσπάθειες είναι ο καταλληλότερος τρόπος να καταπολεμήσουμε τη ρωσική απειλή που πολύ σωστά παρουσιάσατε ή πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από ε, τις ε, χώρες της ανατολικής, που έχουν μια ανατολική οπτική γωνία για την ε, συνολική ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Τι ε, μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Πέτερσεν, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ για αυτή τη διεξοδική παρουσίαση. Πλούσιες ιδέες για τις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα προσυπογράψω στα συμπεράσματά σας ότι πρέπει να επιτύχουμε την Ενεργειακή Ένωση και θα συμφωνήσω και ως προς τη σημασία της. Η ερώτηση μου είναι αν θα μπορούσατε να αναπτύξετε λίγο το θέμα των μέσων. Πώς να επιτύχουμε μια τέτοια πραγματική ένωση στον τομέα αυτό και τι ρόλο προβλέπετε μακροπρόθεσμα να έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διαδραματίσουν εδώ. Και επίσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και αυτό πώς μπορεί να συνδυαστεί. Επίσης, μπορούμε να αποταμιεύσουμε, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να ε, ε, αυξήσουμε την ανεξαρτησία μας. Αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενος και δυσυσυγητής ο κ. Γιάβορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτήν την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Όμως, τι είδους Ενεργειακή Ένωση ε, χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί το χρειαζόμαστε είναι σίγουρο. Και σε σχέση με αυτό που ο κύριος Πέτρεσεν, αρκεί να δημιουργήσουμε μια ε, Ενεργειακή Ένωση που να εντοπίζεται στα ορυκτά, στις ορυκτές πηγές ενέργειας, δηλαδή την ε, παροχή και τον ανεφοδιασμό σε αέριο που σχετίζεται πολλές φορές με την πυρηνική ενέργεια, το πετρέλαιο και επίσης για τη συνολική μας στρατηγική. Αν μέχρι το 2030 πετύχουμε όλους τους στόχους που περιλαμβάνει η σχετική μας στρατηγική, η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πετρέλαιο, το αέριο και το χάλιβα θα αυξηθεί. Αυτή η στρατηγική λοιπόν είναι αποτελεσματική, είναι χρήσιμη εφόσον αυξάνει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις πηγές ενέργειας, ε, τις ορυκτές εντός εισαγωγικών. Και μήπως χρειαζόμαστε μια στρατηγική που να επικεντρώνεται περισσότερο σε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, σε μέτρα που να τονώνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση τους. Πρέπει να περιορίσουμε την ενεργειακή, εξάρτηση της Ευρώπης. Και πρέπει να πω ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι, πώς να το πω, λίγο απογοητευτική ως προς το εξής. Οι περισσότεροι ομιλητές και τα περισσότερα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακρόαση επικεντρώνονται στις ορυκτές πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο, το αέριο και τον αναφοδιασμό μας αυτά και πολύ λίγα βλέπω ότι θα υποθούν για την ενέργεια και αποδοτικότητα και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ενεργειακής Ασφάλειας. Ευχαριστούμε ο κύριο Χάνκερ που είναι και αντιπρόεδρος. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η πιθανότητα εκβιασμού mm. της Ευρώπης δεν είναι κάτι το mm. καινούριο. Εγώ το θυμάμαι στη δεκαετία του 70 και 80 είχαμε τα ίδια από τις χώρες του κόλπου. Και θυμάμαι την αντίδραση του δυτικού κόσμου η οποία ήταν να επιστρατεύσει όλες τις ενεργειακές πηγές, μα όλες πραγματικά για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Εάν δούμε σήμερα την Ευρώπη βλέπουμε πως συμβαίνει κάτι διαφορετικά. Διαφορετικό. Βλέπουμε χώρες που φτιάχνουν νέα πυρηνικά εργοστάσια. Άλλη μεγάλη χώρα κλείνει τα πυρηνικά της εργοστάσια. Άλλες χώρες ε, αγκαλιάζουν το σχιστολιθικό αέριο. Άλλες δεν θέλουν καμία σχέση. Άλλες χώρες ε, αυξάνουν την δυνατότητα παραγωγής άνθρακα, άλλες πάλι όχι. Και αναρωτιέμαι, είναι πραγματικά δυνατόν να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας εάν δεχόμαστε πως κάθε χώρα κάνει, ε, έχει το δικό της ενεργειακό μείγμα. Ευχαριστώ, ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σβέντες Ξέρω πως είστε πάρα πολύ ε, δυνατός σε αυτόν τον τομέα. Η Λιθουανία και τα κράτη-μέλη, ειδικά η Λιθουανία που έφτιαξε αυτό το τερματικό, προσπάθησε να διδαχτεί από τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί αν δείτε τα τελευταία πέντε χρόνια στην προηγούμενη θητεία θα θυμάστε κύριε Πρόεδρε πόσο δύσκολο ήταν για εμάς να επιτύχουμε κάποια πρόοδο στον ενεργειακό τομέα. Προσπαθήσαμε να αναγνωριστούν ε, οι βαλτικές χώρες ως ευάλωτες ε, Υπάρχει κάποια πρόοδος, υπάρχει μια απόφαση παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως ε, πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο ενιαίο τερματικό αλλά ε, η δυνατότητα αυτή από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει το 2030. Αλλά και πάλι βλέπουμε πως λείπουν οι διασυνδέσεις. Οπότε το ερώτημα είναι γιατί δεν μιλάμε για την ανάπτυξη ή μη του, της πυρνικής ενέργειας και βεβαίως πρέπει να δούμε και τις άλλες δυνατότητες καλές οι ανανεώσιμες κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει, αλλά πρέπει να έχουμε και φτηνή ενέργεια που θα μας επιτρέψει να ανταγωνιζόμαστε. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον ομιλητή τι άποψη έχετε για την πυρηνική ενέργεια, για τα δίκτυα ενέργειας, αν πρέπει να ανήκουν σε ένα κράτος μέλος ή όχι, και τι άποψη έχετε για ένα ενιαίο τερματικό υγροποιημένο αερίο στην Βαλτική. Παραδείγματος χάρη ε, είχε ληφθεί απόφαση να χτιστεί ένα τέτοιο θάλασσα, αλλά εκεί πέρα θα πάγωνε. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε πάρα πολύ στο εμπόριο με την Ρωσία ειδικά με βάση τα τελευταία γεγονότα και λογικό αυτό, αλλά σε σχέση με την Ενεργειακή Ένωση περιλαμβάνει και τα 28 κράτη-μέλη, οπότε χώρες σαν τη δική μου, στην Ιρλανδία δηλαδή. Τι ρόλο βλέπετε ειδικά να παίζει το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, για να αποκτήσουμε αυτή την ανεξαρτησία για την οποία μιλάτε. Εάν δεν υπάρχει ε, πράγματι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματι μιλάμε για την εκμετάλλευση του φθηνού αερίου στον ε, κόσμο. Πώς το βλέπετε λοιπόν, τι βλέπετε να συμβαίνει και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, πιθανώς και η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες βεβαίως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να περιμένετε. Άλλη μία ερώτηση. Παρακαλώ. Ο Σκιώδης, εισηγητής μας. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ε, ε, κύριε Σβέτα, ε, ρώτησαν και προηγούμενοι βεβαίως ε, συνάδελφοι για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ενώ αναφερθήκατε στην εγκατάλειψη από την Λιθουανία του προγράμματος για παιδική ενέργεια, ε, ε, δεν έχουμε ε, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση γύρω από αυτόν τον τομέα της ενέργειας και πώς τοποθετήσετε. Το δεύτερο που ήθελα να πω, έχετε αναφερθεί στην απεξάρτηση από τις πολιτικές της Ρωσίας, στην, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του φυσικού αερίου. Και ε, σημειώσατε, ε, μάλιστα δώσετε ένα χαρακτηρισμό για το ευρωπαϊκό Ναμπούκο. Ε, δεν μας προβληματίζει ότι ακόμα και το εγχείρημα του Ναμπούκο θα μιλούμε για εισαγωγή στην Ευρώπη φυσικού αερίου εάν γίνει κατορθωτό να υλοποιηθεί αυτό το έργο από χώρες που υπάρχει μεγάλη πολιτική αστάθεια. Ε, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά η Τουρκία επιδιώκει να εξασφαλίσει φυσικό αέριο από το Ιράν, ενδεχομένω από το Ιράκ, από την ε, περιοχή της Κασπίας Σάλασσας. Άρα μιλούμε για ε, μια ε, εισαγωγή φυσικού αερίου από χώρες που υπάρχει και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μεγάλη πολιτική ασφάλεια. Δεν θα ήταν λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκόψει πλήρως τους δεσμούς από τη Ρωσία και να βάλει τα αυγά της στο ίδιο καλάθι της ενέργειας ε, και αναφέρομαι σε εισαγωγές από ε, περιοχές που είναι ασταθείς και αυτό θα ενδεχομένως να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή ασφάλεια και την τροφοδοσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Παρακαλώ κύριο Σταγιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι θέμα ο ανεφοδιασμός ενέργειας στην Ευρώπη και η κρίση στη σχέση μας με τη Ρωσία έδειξε τις επιπτώσεις και στις τιμές. Υπάρχει όμως και άλλο ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθούμε και η περιοχή της Βορείου Αφρικής. Η Λιβύη είναι ένας μεγάλος ε, ε, μια μεγάλη πηγή ενέργειας και η αστάθεια στην Βόρεια Αφρική έχει δημιουργήσει τριγμούς, ιδίω στη δική μου τη χώρα, την Ιταλία λόγω χάρη. Οπότε, από αυτήν την σκοπιά δεν χρειάζεται και εδώ μια μελέτη αυτού του θέματος, όπως και το μεγάλο θέμα του σχιστολιθικού αερίου. Στην Ευρώπη έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πέραν τη που θα πρέπει να υπάρχει για να γίνει μια σωστή ανάλυση της δυνατότητας να αναχαιτιστούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς το σχιστολιθικό αέριο και εδώ στην Ευρώπη. Θα ήθελα τη γνώμη των προσκεκλημένων μας. Ευχαριστούμε κύριε Χόκμαρκ. Ευχαριστώ ένα πολύ σύντομο, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Διότι όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια, Ιδίως σε αυτούς τους καιρούς, στο νου μας έρχεται κατευθείαν η Ρωσία, ο μεγάλος μας γείτονας. Δεν ε, ε, κουραζόμαστε ποτέ να λέμε ότι όντως πρέπει να ξαναδούμε τις ορυκτές πηγές ενέργειας και τη στρατηγική αναφοδιασμού μας. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει και η μας για το κλίμα, με κάποιους περιορισμούς, με κάποια όρια που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Η ερώτηση λοιπόν είναι Πώς ε, βλέπετε την ευρωπαϊκή εξάρτηση από διαφορετικές, από τις διάφορες μάλλον πηγές ενέργειας, αυτές που έχουμε σήμερα μπροστά μας, που μας επιτρέπουν να είμαστε πιο ανεξάρτητοι σε σχέση με άλλες, όπως την υδροελεκτρική ή την πυρηνική. Οποιαδήποτε αλλαγή ε, στο επίπεδο αυτών των πηγών ενέργειας έχει ε, μεγάλη σημασία ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε οι εξελίξεις στη Γερμανία προς αυτή την κατεύθυνση σημαίνουν ότι γινόμαστε ακόμα περισσότερο εξαρτημένοι από πηγές ενέργειας που δεν έχουμε εδώ. Και πρέπει να τις εισάγουμε. Μορφές ενέργειας τις οποίες πρέπει να εισάγουμε. Τα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλος κανεί να ζητά το λόγο. Παρακαλώ να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι σημαντικές και ευχαρίστως να τα συζητήσουμε. Στην εισήγησή μου ήθελα να θίξω περισσότερα σημεία, αλλά λόγω του περιορισμού του χρόνου δεν μου να το κάνω. Ε, το βασικό μου μήνυμα ήταν το εξής. Ε, ήταν ότι όταν μιλούμε για ενεργειακή στρατηγική και θέλουμε να χαράξουμε, να σχεδιάσουμε μια τέτοια στρατηγική, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν πρέπει να φοβούμαστε να την αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο αυτή την πραγματικότητα. Ιδάλλως θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι στρατηγικές μας δεν θα είναι οι Δεν θα είναι αποτελεσματικές. Το μήνυμα μου λοιπόν ήταν το εξής. Όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια και σχετικά προγράμματα, δεν μπορεί να έχουμε μόνο οικονομικούς στόχους στο μυαλό μας. Σε κάθε ε, στρατηγική, σε κάθε πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στη στρατηγική μας για την ενέργεια, πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη στήριξη περισσότερη προστασία ε, έναντι της πραγματικότητας, η οποία πρέπει να γίνει κατανοητή όσο έχει σήμερα. Όντως, αυτά ήθελα να πω και κυρίως ε, για το κοινοβούλιο, διότι στο κοινοβούλιο μπορεί κανείς να εκφραστεί ελεύθερα. Η στρατηγική τώρα, η στρατηγική είναι καλή, πρέπει να υλοποιηθεί ωστόσο και να αντιμετωπίσουμε και ένα άλλο στοιχείο της πραγματικότητας. Υπηρέτησα στην κυβέρνηση για 20 χρόνια. Ε, υπάρχει πρόβλημα πολιτικής βούλησης, έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Μιλάμε για εσωτερική ενεργειακή αγορά και την ολοκλήρωσή της ως το 2014, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Ε, γιατί πολιτική βούληση. Αυτό λείπει. Δεν λείπει η ενέργεια, δεν λείπουν οι γνώσεις μηχανικής. Ε, είναι οι αποφάσει των πολιτικών που λείπουν. Αυτές μας λείπουν. στρατηγικέ έχουμε, Τι συζητούμε, αλλά πρέπει να ε, ξαναδούμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε από την πραγματικότητα αυτή και να την παραγνωρίζουμε. Βεβαίως, αν δούμε τις συνιστώσεις της στρατηγικής μας. Βεβαίω, δεν έχει να κάνει μόνο με διασυνδέσεις ορυκτών καυσίμων, αέριο, πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα είναι στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν. Τέτοια στρατηγική έχουμε και στη Λιθουανία, αλλά μια στρατηγική που δεν χρησιμοποιείται. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να εξοικονομήσουμε, να κατευθυνθούμε στις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά από ε, μια περιοχή της Ευρώπης που ε, γνωρίζει πολιτικούς τριγμούς ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην πραγματικότητα. Μια χώρα που προσπαθεί να μας επηρεάσει χειριστικά, να θίξει τη χώρα μας και να την ε, θέσει σε συνθήκες ε, επισφαλής. Να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε σημαντικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία που παράγεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ομοσπονδία της Ρωσίας είναι τέσσερις φορές χαμηλότερη από την τιμή της Λιθουανίας. Η... Ο... Οι σταθμοί λοιπόν που παράγουν ηλεκτρισμό στην Λιθουανία από αέριο πρέπει να ανταγωνιστούν τον ηλεκτρισμό που εισάγεται απευθείας από τη Ρωσία όπου και εκεί τον παράγουν από αέριο ε, τον, ε, την ηλεκτρική αυτή ενέργεια αλλά τέσσερις φορές, με τέσσερις φορές χαμηλότερη τιμή. Αυτό προφανώς ε, κλονίζει την εσωτερική ε, ενεργειακή αγορά όλης της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο θέμα ενέργειας, είναι και θέμα οικονομίας, είναι ανταγωνισμού. Ε, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω βεβαίως να το παρουσιάσω και ως δράμα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτή την πραγματικότητα. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή Ένωση που θέλει να δημιουργήσει. Ξέρετε ότι δεν μπορεί μια νυχτή να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι μια διαδικασία που στον ακαδημαϊκό κόσμο ονομάζεται spill over. Δηλαδή ε, η πραγματικότητα μας οδηγεί να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να προχωρήσουμε με την ε, ε, ενεργειακή ε, κατάσταση της Ευρώπης δεν είμαστε πλέον σε θέση να αντιδράσουμε γέρος. Πρέπει όμως να αντιδράσουμε, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα έχοντας υπόψη και τα συμφέροντα, το όφελος των επιμέρους κρατών για το πρωτογενές energy, το συνδυασμό ενεργειακών πηγών. Αν όμως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα να ακολουθηθεί, θα πρέπει να παραμένουμε πιστοί στο πρόγραμμα αυτό. Εάν μιλήσουμε για τον Αμπούκο, ε, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η οικονομική διάσταση του θέματος, αλλά η πολιτική του περισσότερο. Κάποια στιγμή όλοι αποφασίσαμε να το ε, εφαρμόσουμε, ας το κάνουμε λοιπόν. Ε, η συζήτηση περί οικονομικών είναι άλλο πράγμα. Αλλά τέθηκε το εξής ερώτημα πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Να κάνω την εξή παρομοίωση. Κάποιες φορές σε μια συζήτηση, ε, πολλές φορές σε μια συζήτηση λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομεί δυνατότητες ενεργειακές ή διασυνδέσεις για το αέριο που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες. Δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε αυτές. Όμως, στους προπολογισμούς τους, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αφιερώνουν μεγαλύτερα κονδύλια σε στρατιωτικούς σκοπούς. Για ποιο λόγο, ίσως δηλαδή ε, καλύτερο θα ήταν να υπήρχε μία διασύνδεση, ένας αγωγός, αντί για τρεις ε, επιπλέον δεξαμενές ή ένα υποβρύχιο ή ένα αεροσκάφος ή, τρία ή ένα τεθωρακισμένο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να δούμε ε, ότι το βασικό στοιχείο που μας λείπει είναι η ευελιξία. Όσο περισσότερο ευέλικτη είμαι, τόσο καλύτερη. Αυτό αφορά και τις διαθυνδέσεις, την ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG. Βασική διάσταση του θέματος αυτού είναι η ευελιξία. Κάποιος ε, που συμμετέχει σε διεθνεί διαπραγματεύσει, είτε άνθρωπο είτε χώρα, είναι ελεύθερο. Μπορεί να πει όχι. Σήμερα, κάποια κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης δεν είναι σε θέση να πούν όχι σε μερικού παράγοντε ενέργεια. Τι θα πει αυτό. Αυτό θα πει ακριβώ εξάρτηση. Όσο λοιπόν είμαστε, περισσότερο είμαστε ευέλικτοι, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε και περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, βεβαίω πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις, ε, την προέλευση του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού και τις πηγές μας ε, σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια λαμβάνοντα υπόψη την κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ε, περαιτέρω αυστηρά μέτρα του, Παγκόσμιου Οργανισμού για την, ενεργειακή ασφάλεια, για την πυρηνική ασφάλεια. Μετά, ε, βεβαίω, ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα που θέλουμε, το energy mix, πρέπει οι διάφορε χώρε να αποφασίσουν. Ναι, χρειαζόμαστε και την πυρηνική ενέργεια. Οπότε σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Εάν έχουμε μια διαφορετική ε, πολιτική για το κλίμα και θέλουμε να την ε, προωθήσουμε, πρέπει να τη λάβουμε υπόψη σε όλε τι συζητήσει που γίνονται για τη χάραξη πολιτική Και στην συζήτηση για τι πηγέ ενέργεια να μην ξεχνάμε και την πυρηνική που μπορεί να εξυπηρετήσει του σκοπού μα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισηγησή σας και για τις ε, κατανοητικές σας ε, παρατηρήσεις. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά για μας. Και όπως προαναφέρατε, εκπροσωπείτε την η παροχή ανεξαρτήτων συμβουλών. Είστε ένας ανεξάρτητος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κυρίως διότι ο κύριος Βασίλος Μπαρτούσκα που είναι επόμενος ε, ομιλητής εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο την ε, κυβέρνηση της Τσεχίας. Είστε ο ειδικός απεσταλμένος για την ε, ενεργειακή ασφάλεια και εκπροσωπείτε την κυβέρνηση της χώρας. Επομένως είστε επίσημος εκπρόσωπος αυτής. Βεβαίως και εμείς ακούμε όλες τις απόψεις Τώρα έχουμε το πώ βλέπετε εσεί τα πράγματα και τη δική σα εισήγηση. Κάτι το οποίο θα είναι σαν ένα καμπανάκι, ένα ξυπνητήρι, ούτω ώστε να μπορέσουμε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και από Βόρεια Αφρική μέχρι Μέση Ανατολή και Ρωσία να έχουμε ενεργειακή ε, αυτάρκεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Θα διατρέξω πρώτα απ' όλα γρήγορα τα τελευταία πέντε χρόνια να σου πω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ευρώπη και τέλος να πω λίγα λόγια για την κατάσταση του αερίου στην ε, Ουκρανία γιατί πριν από πέντε χρόνια ήμουν α, ακριβώς ο ενδιάμεσος ε, μεταξύ των τριών αυτών μερών. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την ανασκόπηση των τελευταίων πέντε ετών. Το 2009 θα θυμάστε πως για τρεις εβδομάδες είχαμε διακοπή της ροής του φυσικού αερίου προς τα κρατη λόγω ακριβώ της κόντρας ε, Ουκρανίας, Ρωσίας και βεβαίως άνοιξε και ο αγωγός της Κίνας ε, μέσω του που είχε συμφωνηθεί το 2007 και σε 2,5 χρόνια χτίστηκαν 2.500 ε, χιλιόμετρα αγωγού από το Τουρκμενιστάν διαμέσω Καζακστάν προς Κίνα και από τα Σκένδη, Αστάνα, Μπακού και άλλες πρωτεύουσες με ρωτούσαν τι θα κάνει η Ευρώπη και συνειδητοποίησαν ότι η Ευρώπη βέβαια δεν θα φτιάξει κανέναν αγωγό ενώ η Κίνα το έκανε και μετά εξέπνευσε και επισήμως ο Ναμπούκο μετά από λίγα χρόνια. Μετά βέβαια είχαμε την κρίση στη Βόρεια Αφρική που οδήγησε στην αποσύνθεση της Λιβύης ως ε, χώρα που προμήθευε βεβαίως την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Κατά βάση η Λιβύη τώρα ξέρετε είναι μια Σομαλία στη γειτονιά μας. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Αλγερία τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρώπη όταν πεθάνει ο πρόεδρος Μπουτεφλίκα. Γιατί και εκεί είναι κάπως περίεργη η κατάσταση. Είναι προφανές πως η χώρα ε, ε, ξεπέρασε τον εμφύλιο τη δεκαετία του 90 μόνο και μόνο χάρη στο στρατό. Και βεβαίω Ιράκ, Συρία και Ισλαμικό κράτος. Πριν από τρία χρόνια ακούγαμε διάφορες ομιλίες στην Ευρώπη για, για το Ιρακινό Κουρδιστάν ω πηγή φυσικού αερίου. Τώρα δεν τα ακούμε αυτά γιατί είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς αγωγούς όταν γίνεται πόλεμος. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μάχε σε Ιράκ και Συρία για καιρό. Και ξαναρχόμαστε στο 14 με την κρίση του Ιράν που είναι και πολιτικό Και στην Ουκρανία βεβαίως. Βεβαίως ε, βλέπουμε τι, ποια είναι η αντίδραση. Η ολοκλήρωση της αγοράς στη βορειοδυτική ε, Ευρώπη που συμπεριλαμβάνει τη Γερμανία, τον Πενελούξ και τη Γαλλία αλλά καλύπτει και την Βρετανία, Δανία και την Τσεχία επευκαιρία. Βλέπουμε πως η ολοκλήρωση αυτή των αγορών βοηθά. Για τη χώρα μου η ένταξη σε αυτή την ε, γερμανική αγορά σημαίνει πως φέτος ε, οι εταιρείες μας πληρώνουν για φυσικό αέριο τις τιμές ε, Ρότερνταμ, 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ε, τέτοιες τιμές δεν δίνει η Gazprom βεβαίως. Οπότε θεωρώ πως είναι ένα κομμάτι της απάντησης η ε, ενοποίηση της αγοράς και βέβαιως πιο αξιόπιστες χώρες είτε λέγονται Νορβηγία, Καναδάς, Αυστραλία ή είπα είναι και αυτές μια απάντηση αλλά μεγαλύτερη απάντηση είναι βεβαίως στο εσωτερικό και εδώ πέρα δεν υπάρχει μαγική λύση θα υπάρχει λοιπόν μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Κάποιες χώρες ε, οπωσδήποτε θα αναζητήσουν περισσότερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, άλλες θα στραφούν προς ε, άνθρακα. Θα υπάρξουν επίσης τοπικές πηγές γιατί ε, Σήμερα με την ε, βιομάζα και τοπικές πηγές μπορούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητες οντότητες. Η μεγάλη δυσκολία στην Ευρώπη θα είναι πώς θα έχουμε ανεξαρτησία σε μεγάλη κλίμακα. Για μικρά χωριά ή για πόλεις μέχρι 10.000 ατόμων, σήμερα με τις πηγές που έχουμε μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι οι μεγάλες πόλεις και ειδικά βεβαίως ε, μεγάλη οικισμή γιατί είναι και κοινωνικό το ζήτημα, γιατί σήμερα στη χώρα μου και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί κανείς να γίνει αυτάρκης, αν έχει δικό του σπίτι και κάποια λεφτά. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το πληρώσουν αυτό. Και τα κράτη μέλη τι πρέπει να κάνουν. Οπωσδήποτε θα υπάρξει κάποια όθηση για την πυρηνική ενέργεια. Κάποια άλλα κρατημέλη δεν θα το κάνουν, θα στραφούν στο αέριο, το LNG, υδροηλεκτρικά. Για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Νομίζω πως για χρόνια θα υπάρχει αυτή η επικοινομορφία αλλά κάνω αυτή τη δουλειά μόνο 8 χρόνια βεβαίως, οπότε ίσως κάνω λάθος. Έχω διαπιστώσει πάντως πως δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση. Οπωσδήποτε θα ακούσουμε περισσότερα πράγματα για την αλληλεγγύη και θα ήθελα να πω το εξή. Πρώτα ευθύνη και μετά αλληλεγγύη. Είναι καθήκον του κάθε κράτους μέλους να φροντίσει τους πολίτες του. Η εμπειρία της χώρας μου είναι γνωστή. Τη δεκαετία του 90 φτιάξαμε ε, αγωγούς, και έχουμε και ένα συμβόλαιο από την Νορβηγία ήδη και χωρίς να έχουμε πάρα πολλά λεφτά ήδη τότε. Το μεγάλο θέμα σήμερα είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα γιατί το 2009 ήμουν ο αρμόδιος της ε, Τσεχικής Προεδρίας ε, διαπραγματευόμουν τότε με τον ε, Πρωθυπουργό Πούτιν και τον Γιουσένκο και την Αυτογκάζ και την Ασπρόμ. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα πραγματικά θυμίζει πάρα πολύ το 2009. Δύο πράγματα πρέπει να έχετε κατά νου. Το ένα είναι κάτι το φανταστικό. Δεν υπάρχουν μετρητές φυσικού αερίου στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα για 23 χρόνια είναι. Εδώ και 23 χρόνια είναι ανεξάρτητη χώρα η Ουκρανία. Κανείς τους δεν ασχολήθηκε να βάλει μετρητές. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι γίνονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και αντιλαμβάνεστε πως δεν θα καταλάβει παρόν ποτέ απ' έξω το βαθμό της διαφθοράς που συνδέεται με το φυσικό αέριο. Αν θεωρείτε πως οι δισεκατομμυριούχοι στην Ουκρανία έκαναν την περιουσία τη σοκολάτα, τι να σας πω. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως όλες ε, οι ευρωπαϊκές συμβάσεις με την Gazprom έχουν ως σημείο παράδοσης τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημείο εντός της Ένωσης. Κανείς δεν αγοράζει στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Το 2009 ήταν ε, σαφής η θέση μας, είπαμε πως δεν θα πληρώσουμε ε, εμείς λίτρα. Έχουμε συμφωνήσει με την Gazprom να μας φέρει στην Ευρώπη αέριο, το τι θα κάνετε δεν μας ενδιαφέρει. Και ακούσαμε πολύ παρόμοια ποσά ε, για εκβιασμό δηλαδή και από τον κύριο Πούτιν 4,5 δις δολάρια μας ε, ζήτησε και 5, δολάρια, 5 δισεκατομμύρια δολάρια η κυρία ε, Τιμοσέγκο. Ε, και της λέω το... τα 600 εκατομμύρια λέει είναι ΦΠΑ Ουκρανίας. Μάλιστα. Ε, πάρα πολλοί κόσμος στην Κομισιόν για να επιτύχουμε μια συμφωνία και τα έχω ζήσει εγώ το 2009 και πραγματικά εκτιμώ τη δουλειά που έκαναν. Ήταν δύσκολη η συμφωνία και δεν θα κρατήσει. Εάν πιστεύετε πως θα κρατήσει αυτή η συμφωνία μέχρι το Μάρτιο του επομένου έτους, σας έχω άσχημα νέα. Αποδείχτηκε πως μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω και άρα θα μας ζητήσουν παραπάνω και το Ιράν και η Ρωσία. Γιατί έτσι το βλέπουν χώρες, δηλαδή μας θεωρούν χώρες που είμαστε υπεύθυνε εμείς για την ευημερία την ε, δικιά τους. Ε, και Βεβαίω, ε, κανεί Ευρωπαίο πολιτικό δεν θα πει δεν με ενδιαφέρουν οι πολίτε μου στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία ή στην Ουγγαρία ή ακόμα και στη Σερβία. Εμεί δεν το κάνουμε αυτό, να αφήσουμε τον κόσμο να παγώσει το χειμώνα, ενώ άλλες χώρες αδιαφορούν πλήρως για το λαό τους. Κάτι άλλο που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως ο ρόλος της Gazprom άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Πριν από 50 χρόνια η Gazprom ήταν το βασικό εργαλείο πολιτικής. Επί Γέλτσιν ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως η βιομηχανία. Η Rosneft ήταν η δέκατη τέταρτη ε, ε, σε μέγεθος και η μόνη κρατική. Το ίδιο και η Γκάσπρομ. Μην ξεχνάτε πως το αέριο είναι μόνο το 1 πέμπτο των εσόδων των ε, ανθράκων της Ρωσίας. Τα 4 πέμπτα είναι το πετρέλαιο και βεβαίως η Ρωσνέφτα αναλαμβάνοντας την Γιούκος δηλαδή και άλλες εταιρείες που κατέσχισαν. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται τους τελευταίους μήνες, σε μειώνουν τις παραδόσεις σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία. Δεν ανακοινώθηκε και Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία λέξη, είμαστε η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο ακόμα. Και οπωσδήποτε εμείς πρέπει να κάνουμε κουμάντο στην ενέργεια. Αν είναι να μας εκβιάζουν, τότε πρέπει να δούμε το τίμημα του ε, εκβιασμού ως μέρους της απάντησής μας. Και πάρα πολλές απαντήσεις που κάναμε, ανανεώσιμες νέες πηγές, ενέργειας κτλ. ξαφνικά θα μας φαίνονται πολύ φτηνές. Η ενέργεια πλέον δεν είναι καθαρά ενέργεια, ε, οικονομικό ζήτημα. Αυτό, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, ομιλία σας. Ο κύριος Σαουντάργας, ο εισηγητής μας. ευχαριστώ πολύ για την τόσο σαφή σας τοποθέτηση. Από την οπτική γωνία της εξωτερικής πολιτικής είναι σημαντικό να μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση για τις απειλές που επικρέμονται. Να συμφωνήσω όμως να, δω, να, δούμε, να σημειώσω ότι συμφωνείτε και με τον προηγούμενο μιλήτη, ότι πρέπει να έχουμε και την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου προκλήσει. Για άλλη μια φορά λοιπόν, να επαναλάβω την ερώτησή μου που έθεσα και στον προηγούμενο προσκεκλημένο μας. Από τη δική σας τη σκοπιά, επειδή συνεχίζουμε να βλέπουμε τι γίνεται στην ανατολική μας γειτονιά και ο επόμενος χειμώνας θα είναι ένα τεστ κόπωσης για τα συστήματά μας. Η στρατηγική μας δεν θα πρέπει να ε, έχει χρονικό ορίζοντα για ένα χειμώνα, αλλά να θέσει δίτα θεμέλια και την προετοιμασία για, τον, για τους ερχόμενους χειμώνες. Και όπως είπατε, άλλες χώρες, στην Κίνα, στην Κεντρική Ασία, στην ε, Αφρική, ε, συγκεντρώνουν την πολιτική τους βούληση για να ε, λύσουν τέτοια ζητήματα. Τι ε, μαθήματα λοιπόν μπορούμε να αντλήσουμε από τις καταστάσεις αυτές. Πώς να τα συμπεριλάβουμε στην ενεργειακή μας στρατηγική ώστε να έχει μακροπρόθεσμους στόχους, να είναι βιώσιμη και να είναι ένας πραγματικός στυλοβάτης της ενεργειακής πολιτικής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριο Μπό. Ε, για, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, έχω τις εξής ερωτήσεις σε σχέση με την εισηγήσή σας. Πρώτα πρώτα, να είπατε ότι η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να συνδέεται με, με πολλές αναλυτικές λύσεις. Ακριβώς όπως θα πρέπει να ισχύει και για το φυσικό αέριο, ό,τι ισχύει και για το πετρέλαιο. Οπότε θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το θέμα των ε, υποδομών. Άρα θα πρέπει ομένως να έχουμε νέους τερματικούς. Πολύ καλή ιδέα και για πέστε μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στο εγγύς μέλλον και να έχουμε μια παγκόσμια αγορά που λειτουργεί έτσι. Επίσης είδαμε το ότι οι επενδύσεις για την ε, μεταφορά του φυσικού αερίου είτε με τερματικού συγκροπημένου αερίου είτε με αγωγούς ε, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την ε, ζήτηση. Προσφορά είναι πιο μεγάλη από την ευρωπαϊκή ζήτηση. Άρα αυτό πρέπει να δημιουργήσει πιέσεις στο άμεσο μέλλον όσον αφορά την τιμή του φυσικού αερίου. Άρα θα πέσει η τιμή του φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Έχουμε τον κύριο Πέτερσεν που και εκείνο είναι σκιώδης συγγητή. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγγυσή σας και πάρα πολύ με χαροποίησε το ότι τονίσατε το τι θα γίνει με τις εθνικές πολιτικές για τα σχετικά ζητήματα και επίση τι είπατε για τις ανώσιμε πηγές ενέργεια, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τι λύσει που αναζητούμε. Έχω κάτι να ρωτήσω. Πέραν των όσων είπατε. Η πληροφορική και το hacking επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μέχρι ποιο βαθμό όμως. Γιατί και αυτό είναι ένα από τα πολλά δύσκολα προβλήματα όπως μας αναφέρατε. Ο κ. Γιάβο είναι ο επόμενος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Ακούσαμε τα περί πυρηνική ενέργειας και είπαμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια τοπική πηγή ενέργειας. Επίσης θέλω να επαναφέρω το θέμα της επιρροής της ε, Ρωσίας σε αυτόν τον τομέα, ε, ειδικά για Φινλανδία και Ουγγαρία, όπου η Ρωσαντόμ έχει εμπλακεί στις σχετικές επενδύσεις. Επιλάμε για την ε, εξάρτηση όσον αφορά το φυσικό αέριο, το συζητά αυτό ο κόσμος στην Ευρώπη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και την άλλη εξάρτηση που σχετίζεται με ε, την επιρροή της Ρωσατόμ ο πλευράς τεχνολογίας, οικονομίας κλπ. στην πυρηνική αγορά της Ευρώπης. Η Gazprom, η Rosneft επίσης έχουν ανακατευθεί και με τα έργα της ευρωπαϊκής αγοράς. Και δεν είναι τόσο άμεσα έκδηλα τα σημάδια όπως με το να κλείνουν την κάνουλα. Αλλά πάντως ε, ό,τι κάνουν οι Ρώσοι επιδρά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Σας ευχαριστώ. Είμαστε μια ήπειρος με ενεργειακή εξάρτηση. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Επομένως, είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί προμαθευτές ε, ασκούν πολιτική πέραν της Gazprom. Έχουμε και τις ιδιωτικοποιημένες ε, εταιρείε που κάνουν το ίδιο. Και από το Μάιο του 2014 ξέρουμε τι έχει γίνει μια που έχουμε τώρα το ενεργειακό μείγμα που αφορά την κυριαρχία των κρατών μελών. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Υπάρχουν κάποιες ε, αλήθειες, κάποιες αρχές που είναι αμφίβολες. Έχουμε τις σχετικές οδηγίες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, έχουμε ότι το ότι θέλουμε να έχουμε εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τους τερματικούς για τα νοικοκυριά, για την ε, αποθήκευση, την, την, ε, το, το αέριο, θέλουμε να δούμε τι γίνεται και με τα ορυκτά καύσιμα, αλλά Αυτά είναι γνωστά. Τώρα δούμε. Είναι και το θέμα της, του συντονισμού πέραν της ενημέρωσης, της πληροφόρησης όσον αφορά τις συμβάσεις με τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα πει όμως συντονισμός, κάποιο έλεγχος της ασφάλειας για τα νέα προϊόντα. Επομένως, πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει την εξουσία η Κομισιόν να σταματά κάποια έργα ή προγράμματα εάν υπάρχει θέμα κάποιου κυρίαρχου, δεσπόζοντος, πάροχο. Μόνο ψώνιο. Υπάρχει, επομένως, μόνο ένας πελάτης. Οπότε, να και ποιο είναι το πρόβλημα με την ενεργειακή Ένωση. Άρα είναι θέμα συντονισμού και πληροφόρησης. Ο κύριος Μάνκας, ευχαριστώ πρόεδρε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Βέντας είπε πως σέβεται οπωσδήποτε το ότι κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει ποιο θα είναι το ενεργειακό της ε, μείγμα. Τα κ. Πάντουσκα ε, μας είπε πως ε, αποφάσισαν προσφάτως οι Γερμανοί να απομακρυνθούν από την πυρηνική ενέργεια. Όταν ε, μεγάλες χώρες λαμβάνουν από τη μια μέρα στην άλλη τέτοιες αποφάσεις, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις και σε άλλες χώρες, οπότε θα πρέπει να ενημερώνονται οι, ε, οι χώρες και να συντονίζονται. Ε, το δεύτερο μου ερώτημα αφορά το εξής τις πηγές ενέργειας οι οποίες είναι κάπως ε, ας πούμε ανασφαλής. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τούσκ για μια κοινή πολιτική αγοράς ενέργειας και έτσι επανερχόμαστε βεβαίως στο ζήτημα της ε, κοινής προμήθειας πρώτων υλών. Σας ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει να δω πώς βλέπετε την οικονομική κατάσταση της Ρωσίας. Ήδη πριν από την οικονομική κρίση υπήρξε δραματική ε, επιδείνωση της κατάστασης και βεβαίως ενδιαμέσως καταστράφηκε και αρκετή πίστη στην ε, ρωσική οικονομία. Τι επίδραση ότι θα έχει αυτό στην ε, προμήθεια ενέργεια. Σας ευχαριστώ κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπερασπιστώ την ε, καγκελάριό μου που πολλοί λένε πως βιάστηκε στην απόφαση για την απομάκρυνση από την πυρηνική ενέργεια. Είναι λάθος αυτό. Το συζητάμε εδώ και 30 χρόνια στη χώρα μου και η απόφαση της κυβέρνησης ε, νομίζω ε, τη στηρίζουν αυτή τη στιγμή πάνω από 85% των Γερμανών και όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Τρεις ερωτήσεις προς τον κύριο και Σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Πρώτον, αναφέρθηκε ήδη πώς οι δυνατότητες ε, ε, LNG είναι αυτή τη στιγμή πάνω από την χρήση. Θεωρείτε λοιπόν πως χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις εκεί και ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τα επόμενα πέντε με 10 χρόνια για πιθανές εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ. Αναμένεται να υπάρξει εκεί πέρα κάποια συνεισφορά για την ευρωπαϊκή ενέργεια. Μετά αναφέρεται το ζήτημα της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Θεωρείται πως οι στόχοι της πρόσφατης συνόδου κορυφής είναι αρκετά φιλόδοξοι για να ενισχύσουν την ανεξαρτησία μας. Και τρίτον, όσον αφορά την ζωτική, ε, τις ζωτικές υποδομές ενέργειας. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ έχουν πάρα πολλά μέσα νομικά για να υπερασπίσουν τις ζωτικές ενεργειακές υποδομές απέναντι σε παρεμβολή από τρίτες χώρες που πηγαίνουν πολύ παραπέρα από τα δικά μας μέσα. Θεωρείτε πως θα πρέπει να έχουμε κάποια περισσότερα εργαλεία στην ε, διάθεσή μας. Ευχαριστώ ο Σκάιντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ειδικά αυτά τα οποία αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις του 2009 να σκεφτούμε λίγο την ε, ενεργειακή ανεξαρτησία. Φαίνεται πως υπάρχουν δύο είδη ανεξαρτησίας. Η μία είναι ε, πλήρης ανεξαρτησία από εισαγόμενες πηγές. Να σκεφτούμε π.χ. μια αγορά σαν της ΕΠΑ. Αν δεν κάνω λάθος από το πετρελαϊκό εμπάργο στα τέλη δεκαετίας του 70 είχαν θέσει ως στόχο να γίνουν ανεξάρτητες. Ε, κανείς δεν το πίστευε, αλλά τώρα τα κατάφεραν με το σχιστοελιστικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν βασίζονται πλέον στις αγωγές, έχουν γίνει εξαγωγείς. Κάτι το οποίο δεν θα το πιστεύαμε πριν από πέντε χρόνια. Θεωρείτε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε καθόλου εισαγωγές ή η ανεξαρτησία που μιλάτε είναι να έχουμε τη δυνατότητα να λέμε, είναι να έχουμε τη δυνατότητα να λέμε όχι σε κάποιον ε, πιθανό προμηθευτή γιατί ε, έχουμε πολλούς άλλους προμηθευτές για να πούμε σε οποιονδήποτε έναν από αυτούς ένα όχι. Σας ευχαριστώ κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ. Για μένα η κρίση του αερίου είναι κρίση θέρμανσης, οπότε είναι πραγματικά έκπληξη πως ε, η απάντηση είναι να αλλάξουμε και άλλο τις πηγές. Ε, καταναλώνουμε λιγότερο ε, φυσικό αέριο γιατί, γιατί έχει καταρρεύσει το ETS και δουλεύουν στο full τα εργοστάσια άνθρακα. Νομίζω πως ε, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που είχαν ποτέ. Οπότε, οπότε η κρίση του φυσικού αερίου είναι μια κρίση θέρμανσης στην Ανατολική Ευρώπη. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για το τι θα κάνουμε για την θέρμανση, να φύγει το φυσικό αέριο από τη θέρμανση. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εγώ τα βλέπω έτσι μετά την επανάσταση στην Ανατολική Ευρώπη, υπήρχε ένα γενικό ξεπούλημα όλων των περισσιακών στοιχείων στους πολίτες. Οπότε στην Ανατολική Ευρώπη ε, είναι πολύ μεγαλύτερη η ιδιοκατοίκηση, αλλά μου λένε πως 60% των Ανατολικοευρωπαίων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κτίρια που δεν είναι σωστά μονομένα και δεν έχουν λεφτά να τα μονώσουν. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και μετά, για κάτι το οποίο σωστά έθεσε ο κύριος Λεβαντόφσκι. Κάτι λυπηρό στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον συντονισμό της Ευρώπης. Ε, το κείμενο αυτό νερώθηκε και πλέον έχει φτάσει να μην έχει κανένα νόημα. Και βεβαίως εδώ πέρα οφείλουμε να κατηγορήσουμε την ε, Γερμανία αλλά και η Πολωνία δεν αντιστάθηκε παρά τα λόγια ότι θα δώσει τη μάχη στο Συμβούλιο. Οπότε το πραγματικό ζήτημα είναι ο συντονισμός. Έχουμε την ευκαιρία να, να διαπραγματευτούμε τα δύο τρίτα των ε, συμβάσεων φυσικού αερίου τα επόμενα 8 χρόνια. Από την υπηρεσία ενέργειας είναι αυτά. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία λοιπόν. Αλλά αυτό μόνο εάν βοηθήσουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας για το ζήτημα αυτό του καλύτερου συντονισμού. Και τελευταίο ερώτημα. Οι, αγορα... συμφωνίες αγοράς φυσικού αερίου. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός για την ιδέα κοινή ε, αγοράς ε, γιατί η αντίδραση από την άλλη πλευρά θα είναι καρτέλ των πολιτών. Οπότε τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε. Ε, συνάδελφοι, είπαμε δύο λεπτά ο καθένας. μισή λεπτά εντάξει αλλά όχι τρία. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να στηρίξω στον άλφο τον κύριο Μπιουτικόφερ, γιατί από όταν έκλεισε τα πυρηνικά εργοστάσια η Γερμανία δεν λείπει ενέργεια. Αντιθέτως παράγουμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι πριν. Και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όσον αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία. Επίσης θα με ενδιέφερε ποιες είναι οι προτάσεις του Συμβουλίου γιατί εγώ περίμενα κάτι το πιο φιλόδοξο, ίσως έχετε κάτι να μας πείτε για την ενεργειακή ασφάλεια και ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει μια πρόταση από την Πολωνία για να υπάρξει ακριβώς μια κεντρική ε, προμήθεια και ίσως μια ανάλογη υπηρεσία με την Ευρατόμ ή κάτι άλλο, μια εθελοντική κοινοπραξία που θα αναλάβει αυτή τη δουλειά. Θα ήθελα να μάθω την άποψή σας επ' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Mm. Ο κύριος Γιάνκεβιτς, ευχαριστώ πρόεδρε. Έγινε μια ευρεία συζήτηση τους τελευταίους μήνες για τα θέματα αυτά και ε, ευτυχώς διότι η κατάσταση στην εξωτερική πολιτική και διεθνώς είναι ε, κρίσιμη με την κατάσταση στην Ουκρανία. Αλλά και απόψεις της κοινή γνώμη είναι σημαντικές για την όλη συζήτηση. Δηλαδή οι εντάσεις στην Ομοσπονδία της Ρωσίας και οι τεταμένες μας σχέσεις μαζί τους είναι ένα θέμα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κύριε Μπαρτούσκα. Ε, η ενεργειακή μας ασφάλεια θα πρέπει να περιοριστεί, να βασιστεί στην, στον περιορισμό της εξάρτησης από τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Gazprom. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι συστημικοί παράγοντες, όπως η περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, λόγω χάρη. Ε, αυτή την άποψη την έχουν υποστηρίξει πολύ ε, ψηλά ιστάμενοι μεταξύ των οποίων και πολλοί επίτροποι. Εγώ δεν την πιστεύω την άποψη αυτή. Εάν περιορίσουμε τον ανεφοδιασμό μας από το ρωσικό αέριο δεν θα καλύψουμε απλώς το ε, ενεργειακό κενό που έχουμε με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν είναι αυτή η λύση για την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή μιλούν για την ανάγκη να απαλλαγούμε και να ε, περιορίσουμε τη χρήση χάλιβα οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολιτικοί ή μιλούν πολύ για το σχιστολιθικό αέριο αντί να στηρίξουν τις πηγές ενέργειας που είναι τελείως ανεξάρτητες. Μιλούν λοιπόν για την ε, απαλλαγή Απεξάρτηση από τον άνθρακα. Εσείς κύριε Μπαρτούσκα τι άποψη έχετε. Ε, αυτή η απεξάρτηση είναι μια σωστή κατεύθυνση. Θα λύσει τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ο Ισκιώδης εισηγητής ο κύριος Ταμπουράνο. Η ερώτησή μου είναι περισσότερο διευκρινιστική. Διότι υπάρχει ένας μύθος για την αμερικανική ενεργειακή ανεξαρτησία οι οποίες το 2013 το 11% της ε, κατανάλωσης αερίου τα, την ε, εισήγαγαν. Το εισήγαγαν με, 9,6 βαρέλια πετρελαίου από, παράγοντα, από παράγωγα ε, μέχρι το 2016. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν με τι στοιχεία οι περισσότεροι από εμά λένε ότι έχουν φτάσει την ενεργειακή ανεξαρτησία οι Αμερικανοί. Κάτι που βασίζεται σε στοιχεία που εύκολα μπορεί κανείς να εξακριβώσει από τις εφημερίδες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο λοιπόν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχουν ε, άλλα αιτήματα. Να προσθέσω και εγώ σε συνέχεια όσων είπαν ε, ο κ. Λεπαντόφσκι και ο κ. Τούρμες ότι κατά την άποψή μας η ενεργειακή κοινότητα ήταν μια δημοφιλής ιδέα αλλά το δύσκολο ήταν να τα εξηγήσουμε όλα αυτά στα κράτη-μέλη και να τα υλοποιήσουν. Διότι προσπαθήσαμε με επιμέρους επισκέψεις να την ε, προωθήσουμε την ενεργειακή κοινότητα. Χρειάζεται κοινή ε, πρικοδότηση της ενεργειακής αυτής ε, προσπάθειας. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για την Ενεργειακή Ένωση. Ήταν ε, εύκολο να λάβουμε κάποιες νομοθετικές αποφάσεις, αλλά επιτέλους πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα. Κοινές αγορές θα οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ή καθόλου. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ειδικέ αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε κατευθείαν. Και το σχολίασαν κι άλλοι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο. Δώσατε πέντε λεπτά, Πρόεδρε, οπότε θα είμαι πολύ σύντομο. Για τις αγορές αερίου. Είτε θα δημιουργήσουμε μια χώρα ισβαρος κάποια έργης ευρωπαϊκή αγορά και κανείς ε, πάροχος δεν θα εκβιάζει μια χώρα εις βάρος κάποιες άλλες ή υπέρ κάποιες άλλες. Εάν δείτε τι γίνεται στη γερμανική αγορά και αλλού έχουμε 18 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ανά μεγαβατόρα. Δηλαδή τα μισά από όσα πληρώνει η Λετωνία για το αέριό τη που αναφοδιάζεται στην ε, Ρωσία. Εμείς πληρώνουμε περισσότερα από ό,τι λόγω χάρη η Σλοβακία. Ε, άρα δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προβλέψουμε μια κοινή αγορά αέριου για όλες τις εταιρείε. Δεν το νομίζω. Τώρα, για το hacking και τα εφή δίκτυα. Αυτό είναι Κάτι πολύ ε, σημαντικό. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο διαδίκτυο, για να το πω έτσι με μια παρομοίωση, για την ενέργεια. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε και την προστασία μας, διότι εάν έχει κανείς περιφραγμένο σπίτι με εσωτερική παροχή ενέργειας, μπορεί να είναι αρκετά ανεξάρτητος αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι αυτό εφικτό. Τώρα για την ε, ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ενέργεια και την ε, κυριαρχία των, ε, την αυτάρκεια των κρατών μελών. Αυτό ήταν κάτι που ανέκαθεν η Ευρώπη το ε, καλλιεργούσε. Ε, ήμασταν πάντα τα κυρίαρχα εθνικά κράτη. Δεν μπορούμε να γίνουμε μεγάλη σαν την Κίνα και να λύνουμε τα προβλήματά μα έτσι. Και οι περισσότεροι πολίτε μα νομίζω κάτι τέτοιο επιδιώκουν τώρα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Από την άνθηση του σχιστολιθικού αερίου το 2008 ε, και 2009 δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα γιατί θα είχαμε εισάγει υγροποιημένο αέριο εάν δεν είχαν την τον εσωτερικό τους ανεφοδιασμό οι Ηνωμένε Πολιτείε. Για έκτη συνεχή χρονιά λοιπόν έχουν πέσει οι τιμές του υγροποιημένου αερίου και υπάρχει σοβαρή πίεση εσωτερικός για να διατηρήσουμε αυτό το πλέον έκτημα ε, στην Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο θέμα στι Ηνωμένε Πολιτείε για την ανεξαρτησία τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία λεπτομέρεια. Πολύ ωραία απεικονίσατε την πραγματικότητα, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητε ω προς το ακατέργαστο πετρέλαιο. Όμω στο είμαι ακατέργαστο, σε κάποιε πολιτείε είναι πολύ, στο αργό πετρέλαιο είναι πολύ λιγότερο ε, ανεξάρτητα σε συγκεκριμένα σημεία όπως η Λιουιζιάννα. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό για όλες τις ε, χώρες. Δεν μπορεί καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απολύτως ανεξάρτητη Για την ανεπεξάρτηση από το Χάλιβα ήταν μια πολύ καλή παρατήρηση, αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να δούμε το αέριο ως εμπορικό αγαθό. Την θέρμανση μπορούμε να την κάνουμε με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με ξύλο, με χάλιβα, με συγκεκριμένες υποδομές και εγκαταστάσεις. Αλλά δείτε πόσες ε, σόμπες πουλήθηκαν κάτω στην Ανατολική Ευρώπη, σόμπες που κινούνται με αέριο και θερμάστρες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Εάν ε, βασιζόσασταν πλήρω στο αέριο, αυτά θα τα βλέπατε διαφορετικά. Δηλαδή, το θέμα είναι πώ αντιδρούν και οι ίδιοι πολίτε και οι τοπικέ κοινότητε. Δεν αρκεί μόνο οι κυβερνήσει να πιέζουν του πολίτε να αλλάξουν τη συμπεριφορά του. Όταν ακούνε όλοι Gazprom, ε, δρυμής χειμώνας, ε, πώς θα το... και ακούνε ότι πρέπει να προετοιμαστούν. Πώς να προετοιμαστούν χωρίς αέριο. Και ας είμαι λίγο ασύνδεξος προς το τέλος. Είμαστε ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο και μια από τι πλουσιότερες επίρους. Α χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις που έχουμε για να κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη και ίσως και τις χώρες που εξάγουν προς εμάς, ας τις δυσκολέψουμε λίγο τη ζωή. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την εισήγησή σας, αλλά και για τις απαντήσεις που δώσατε. Και τώρα, ας επανέλθουμε. Έχουμε τον καθηγητή ο Κομπάρντι από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Θα μας πει τώρα για τα ορυκτά κάψιμα, τους ορυκτούς υδρογονάνθρακες και όσον αφορά επίσης τα ε, αποτελέσματα επί των ε, μειωμένων αποδόσεων, της μειωμένης αποδόσεως της Κομπάρντι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω σε ένα τόσο ε, ε, εξαιρετικό ακροατήριο στο Ίδρυμα στο Ινστιτούτο για την ε, Χημεία ε, στο οποίο εργάζομαι θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα απορίσματα της δουλειάς μου στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Σήμερα θα επικεντρωθώ στο πετρέλαιο, αν και μιλάτε πιο πολύ για το αέριο και όλοι γνωρίζετε τι κρίση ε, προκύπτει τους τελευταίους μήνες, έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια νέα ε, κρίση ε, για το αργό με το αργό πετρέλαιο και την μείωση των τιμών, κάτι που είναι εξίσου αρνητικό για την αγορά με την αύξηση των τιμών μπορεί να νομίζετε ότι οι τιμέ του πετρελαίου, οι χαμηλέ τιμέ είναι κάτι το καλό, αλλά δεν είναι έτσι γιατί δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνουν, όπως θα προσπάθησα να σας αποδείξω. Για να δούμε τα πράγματα λοιπόν υπό μια προοπτική να σκεφτούμε λίγο το ιστορικό των τιμών του πετρελαίου. Και θα πάμε πίσω περίπου έναν αιώνα, 80 χρόνια. Όπως βλέπετε, η κόκκινη γραμμή, παρουσιάζει τις τιμές με τη διόρθωση του πληθωρισμού και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια όρια. Δεν μπορούν να πάνε πολύ ψηλά οι τιμές, διότι αν συμβεί αυτό δεν μπορούν πλέον οι άνθρωποι να αγοράσουν πετρέλαιο. Οπότε έτσι ε, την, με υποοικονομικούς όρους καταστρέφεται η προσφορά η ζήτηση μάλλον. Επίσης, αν είναι πολύ χαμηλέ οι τιμέ, οι πετρελαϊκές εταιρείε δεν μπορούν να παράγουν και να έχουν κερδοφορία. Οπότε δεν παράγουν. Κανείς δεν πουλά με ζημία. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και τα τελευταία χρόνια είχαμε με τέτοια τάση στις τιμές του πετρελαίου. που είχαν αυξητική τάση. Αφού όμως υπάρχει αυτή η τάση στην αύξηση, ε, πρέπει να λάβουμε φυσικά τις υπόλοιπες τάσεις. Γιατί ήταν τόσο υψηλές οι τιμές ε, του πετρελαίου, δεν τις επιβάλλει η Goldman Sachs. Έχουμε φτάσει την κερδοφορία στις Ηνωμένε Πολιτείες 120 ε, δολάρια ανά βαρέλι. Δηλαδή με το σχιστολιθικό αέριο, ε, το σχιστολιθικό αέριο, τον ε, πισούχο ε, σχιστόλιθο που είναι διαφορετικά πράγματα, ξεπερνάμε τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά μόνο έτσι μπορεί να είναι κερδοφόρα αυτή η παραγωγή. Με τέτοιες τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα. Αν δεν είναι σε αυτό το ύψος οι τιμές, Τώρα, αν δείτε που έχουν φτάσει οι τιμέ, πριν 5 λεπτά τι κοίταξα, έχουν κατέβει από τα 57 δολάρια το βαρέλι. Πώ θα κάνετε κανεί παραγωγή κατά αυτόν τον τρόπο, πώ θα ξοδέψει χρήματα για τέτοιου είδου παραγωγή, θα πουλάει με ζημιά. Και στα αριστερά βλέπετε μία εκτίμηση του κόστους παραγωγής πετρελαίου, ενώ στα δεξιά βλέπετε πώς, σε τι τιμή πωλείται το πετρέλαιο. Είναι κάπως ε, ξεπερασμένη ίδια αριθμή, είναι από την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει και άλλη ε, πτώση στις τιμές. Έχουμε φτάσει τα 76 δολάρια το βαρέλι χοντρικά σήμερα. Όπως βλέπετε, οι τιμές αυτή τη στιγμή 76 δολάρια το βαρέλι αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των ε, περιοχών που παράγουν πετρέλαιο. Εάν μείνουν εκεί οι τιμέ, θα πρέπει να μειώσουμε κατά 10% την παραγωγή μας. Εάν υποχωρήσουν κι άλλο, θα πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδα που μας φαίνονταν φυσικά πριν από 10 χρόνια. Αλλά εκεί θα χάσουμε 50% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η τάση, τι προκαλεί αυτή τη συμπεριφορά. Το πρόβλημα είναι πολύ απλά ότι η παραγωγή πετρελαίου κοστίζει περισσότερο όλο και περισσότερο. Για τον εξή απλό λόγο, κάτι που ονομάζω ε, την εξάντληση του πετρελαίου. Δηλαδή, το φτηνό πετρέλαιο έχει ήδη παραχθεί. Τώρα πρέπει να περάσουμε στις ακριβότερες μορφές ε, παραγωγής. Αυτή είναι η τάση στην παραγωγή παγκοσμίω και βλέπει κανείς το γαλάζιο κομμάτι του γραφήματος. Εδώ βρίσκουμε το, τη σύνθεση στην παραγωγή η οποία είναι σταθερή τα τελευταία δέκα χρόνια. Όμως, λόγω του κιτρίνου και του μαύρου κομματιού, ε, έχει αυξηθεί η παραγωγή. Εκεί έχουμε το αμερικανικό και καναδέζικο σχιστολιθικό πετρέλαιο. Οπότε μπορεί κανείς να αυξήσει την παραγωγή του πετρελαίου του χρησιμοποιώντας ακριβότερες πηγές, ακριβότερους τρόπους παραγωγής. Αυτό που εκπροσωπούν οι σημερινές Συζητάμε πάρα πολύ τον πισούχο σχιστόλιθο και το σχιστολιθικό αέριο που είναι πολύ κοντινά. Ε, βλέπετε εδώ αυτό το κομμάτι σχιστόλιθου, ένα κομμάτι πέτρας, πετρώματος, από το οποίο παράγουμε και το σχιστολιθικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο. Δεν είναι απλό δεν αρκεί κανεί να ανοίξει μια τρύπα στο έδαφο. Πρέπει να γίνει υδρορογμάτωση. Πρέπει να διασπαστεί το κομμάτι αυτό πετρώματο. Υπάρχουν πολλέ τεχνολογικέ ε, μέθοδοι που πρέπει να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα. είναι πανάκριβε. Είναι πολύ όμορφε ε, οι τεχνολογικέ λύσει. Ε, βλέπετε αυτό το κινητό που κρατάω ότι ωραίο γκάτζετ είναι, αλλά δεν μπορεί κανεί να σπάσει αυτό το πέτρωμα χρησιμοποιώντα το τηλέφωνο. Το είδο τη τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ακριβό. Και ο ακριβότατος αυτός ε, εξοπλισμός με αυτή την ταχύτατη πτώση στις τιμές του σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού ε, πετρελαίου ε, είναι καταπληκτικός. 80% πτώση τα τελευταία τριετία είχαμε και πρέπει να συνεχιστεί η υδρορογμάτωση. δηλαδή, με πολύ υψηλό κόστος πρέπει να καλυφθούμε από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αλλά οι τιμές δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την κάλυψη. Οπότε το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μπορεί να τροφοδοτήσει αυτή την παραγωγή και η παραγωγή θα πέσει. Αυτό ε, το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στην παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίω υπάρχει αυτή η γενικευμένη ανησυχία αν συνεχίσει η πτώση των τιμών θα υπάρξει και η πτώση στην παραγωγή. Αυτό θα επηρεάσει τους πάντες και την βιομηχανία και τον κλάδο και εμάς που είμαστε οι καταναλωτές, οι τελικοί πελάτες ε, και ε, αποδέκτες της παραγωγής. Πέρα από το υψηλό κόστος όμως υπάρχει το γεγονός ότι χρειάζεται και ενέργεια για να ε, παραχθεί ενέργεια. Δηλαδή για να σπάσουμε από το πέτρωμα, για να γίνει η υδρορογμάτωση λεγόμενη πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενέργεια. Με μια αναλογία που διαρκώς μειώνεται τον τελευταίο αιώνα βεβαίως στην αρχή ε, η αναλογία ήταν 1 προς 100 για το σημαντικό πετρέλαιο. Τώρα είμαστε περίπου στο 10-15, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς 1 για να παράξει 15. Όταν μιλάμε για το σχιστόλι θα είμαστε κάτω από το 10. Οπότε ο παράγοντας αυτός, ο παράγοντας της... Ε, της των κοιτασμάτων είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτική αντίδραση. Να σας δείξω εδώ ένα διάγραμμα για, τις, ε, για τα αποτελέσματα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών βλέπετε ότι τα, οι ανανεώσιμες πηγές αυτή τη στιγμή σήμερα σε υπό συγκεκριμένε συνθήκες μπορούν να συγκριθούν με το πετρέλαιο, δηλαδή ως προς την παραγωγή ενέργειας. Εάν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει τις ανανεώσιμες για να παράξει πετρέλαιο, δηλαδή για καύσιμο για την παραγωγή πετρελαίου, είναι άλλο πράγμα. Όμως βλέπετε ότι η απόδοση ε, αυξάνεται, διότι ε, βελτιώνεται και η τεχνολογία. Και αυτό διότι υπάρχει εξάντληση γενικότερα. Οπότε αφού περιορίζονται τα ορυκτά καύσιμα ε, και συνεχώς μειώνονται, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί στο μέλλον και θα στραφούμε περισσότερο στις ανανεώσιμες. Σας δείχνω εδώ ένα διάγραμμα για το τι γίνεται και με τις επενδύσεις, διότι οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να μας δώσουν ενέργεια, αλλά πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις από αυτό το τομέα, εάν θέλουμε κάτι να πετύχουμε. Να ολοκληρώσω τώρα, διότι με έχει τρομοκρατήσει ο συντονιστής εδώ ότι πρέπει να παραμείνω στα 10 λεπτά. Ε, γιατί για την παραγωγή ενέργειας χρειάζεται ενέργεια. Η, παρα όχι λόγω οικονομικών ή πολιτικών παραγόντων, αλλά λόγω της εξάντλησης μειώνεται η παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Οι υψηλές τιμές καταστρέφουν τη ζήτηση, οι πολύ χαμηλές τιμές καταστρέφουν την προσφορά. Είναι μια κατάσταση περίπλοκη από την οποία μας πρέπει να ξεφύγουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι πολιτικές συζητήσεις που γίνονται για την ενεργική ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η μόνη δυνατότητα που έχουμε για να πετύχουμε την ενεργειακή αυτάρκεια είναι να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές και να ε, ακολουθήσουμε το δρόμο που έχει επιλέξει η Ευρώπη για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών. Ένα σημαντικό τμήμα του ενεργειακού μίξ που θέλει να πετύχει. Σας ευχαριστώ και εδώ υπάρχουν τα στοιχεία ε, στο διαδίκτυο εφόσον σας ενδιαφέρουν σε, αυτό το, σε αυτή τη σελίδα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ε, ομιλία σας. Κύριε Σαντάργας, το λόγο ως εισηγητής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν αυτά πάρα πολύ σαφή, ήταν η ανάλυση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με το τι συμβαίνει στις ε, αγορές του πετρελαίου. Πάρα πολύ σημαντικό, μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τέτοια εξάρτηση ε, από τις εισαγωγές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στο τέλος και σε, ότι είναι σημαντικό ότι είπατε σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής. Συμφωνώ. Πάντως, τώρα θα ήθελα να δούμε κάτι σχετικά με το σημερινό μας ε, θέμα. Μια που είστε ένας εμπειρογνώμονας στα θέματα και στην ε, διαδικασία παραγωγής του πετρελαίου και μας ε, αποκαλύψατε το τι γίνεται, τι θα γίνει μακροπρόθεσμα και τι, πώς έχουμε αυτές τις ε, βραδίες τάσεις εξέλιξης των της τεχνολογίας που μπορεί να είναι βιώσιμες αλλά είναι αργές και έχουμε επίσης και αυτού του είδους τις απότομες βίες διακυμάνσεις των τιμών και έχουμε κάποιους περίπλοκους μηχανισμούς, έχει να κάνει αυτό και με την κρίση, αλλά κατά τη γνώμη σας, κατά τη γνώμη σας, ποια πολιτικά γεγονότα, πώς η γεωπολιτική κατάσταση επηρεάζει τις τιμές ή την τιμή του πετρελαίου, από δική σας οπτικής γωνίας, τι λέτε, μπας και έχουμε τώρα ένα μέσον για ρύθμιση, για χειραγώγηση ε, των τιμών ε, κάποιες μεταβολές που έχουν σχέση με την οικονομία. Συμφωνώ. Λέει ο κύριος Έριξον με τα περισσότερα τα, από όσα μας είπατε σχέση με το πώς εξελίσσονται τώρα τα πράγματα και το τι θα πρέπει να κάνουμε ε, στο μέλλον από πλευρά Ευρώπης, τόσο ώστε να ανταποκριθούμε στην κατάσταση και θα ήθελα να μου εξηγήσετε Πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση, μήπως επίσης έχουμε κάποιο είδους πόλεμο αγοράς ή αγορών. Έχουμε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στη ΣΥΠΑ. Παράγουν πολύ περισσότερο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο εκεί, οπότε πένσορο ορυκτά καύσιμα ρίχνουν στην αγορά. Βλέπουμε τις αντιδράσεις της Σαουδικής Αραβίας περισσότερη, μεγαλύτερη παραγωγή τώρα από ό,τι πριν, γιατί χάνουν θέσεις στην αγορά, τιμήματα της αγοράς. Πέφτουν οι τιμές. Κατακριμνίζονται ταχείες, οπότε να. Τα αποτελέσματα αυτού του πόλεμου στην αγορά η Σαουδική Αραβία θέλει να φρενάρει κάποιες από τις ακριβές επενδύσεις. Ιδίως για Καναδά και ΙΠΑ. Αυτό δεν είναι ένα κομμάτι της πίτας στο οποίο αναφερθήκατε. Ο άλλος και ο δισηγητής, ο κύριος Γιάμπορ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με μεγάλη ικανοποίηση. Άκουσα, εδώ, εδώ είμαι, λέει ο κύριος Γιάμπορ. Μεγάλη ικανοποίηση άκουσα την εισήγησή σας και θεωρώ ότι πραγματικά μας ε, εξηγήσατε τις στρατηγικές πτυχές των ενεργειακών θεμάτων τι γίνεται με τη Ρωσία, τι γίνεται με την Ουκρανία, με το φυσικό αέριο, με την προμήθεια για το χειμώνα προς την Ευρώπη και έχουμε τώρα μια εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια ή και δεκαετία η αγορά. Τι γίνεται με τα καύσιμα, τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση. γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω τεχνολογίας γίνονται όλο ένα και φτηνότερες και ανταγωνίζονται όλο ένα και πιο δυνατά τα, τα καύσιμα ήδη. Σας ερωτώ, δεδομένης αυτής της καταστάσεως, γιατί είναι από το πρόβλημα που έχουμε για την στρατηγική ε, της ενεργειακής ασφάλειας, είναι πραγματικά μια στρατηγική δεν είναι το θέμα το να δούμε το πώς θα δώσουμε τη μάχη για την ενεργειακή ασφάλεια μακροπρόθεσμα ή μήπω ε, είναι το θέμα του πώς θα έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για τον επόμενο μήνα ή για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Επίσης, για πέστε μας, ένα από τα βασικά βήματα που θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια είναι το πώς θα μπορέσει να έχει κάποιους μακρόπνοη ε, ενεργειακή ασφάλεια. Για να δούμε επομένω πώ θα μπορέσουμε στι ανώσιμε πηγέ να επενδύσουμε στην ενεργειακή αποδοτικότητα και να δούμε πώ τελικά θα είμαι ει θέση να εξασφαλίσουμε αυτή την ενεργειακή ασφάλεια για την ε, Ευρώπη και να στραφούμε ε, μακριά από αυτή τη, τη, τη, στενή οπτική τη εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και σκουέρια κλπ. Ο επόμενο. Κένετε. Yes, thank you very much. Ο κύριο Κέλλη, ο Σκέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά όσον αφορά τη διαμόρφωση τη τιμή του πετρελαίου, αλλά για πετε μα, ισχύει δεν ισχύει ότι τα κέρδη έχουν συρρυκνωθεί, αλλά η ζήτηση παραμένει και θα παραμείνει εκεί που είναι και ότι άπαξ και είναι κερδοφόρα η παραγωγή άντλης του πετρελαίου, όσο και να έχει πέσει η ζήτηση, όσο και αν πέσει. Και επίση για πετε μα τώρα με το ε, πετρέλαιο. Είδατε τι πριν από κάνα δύο χρόνια. Είχαμε επένδυση η οποία είναι τόσο μεγάλη που δεν πρόκειται να μειωθεί η παραγωγική δυνατότητα της ε, παραγωγής πετρελαίου από το σχιστόλιθο στο ορατό μέλλον. Επίσης, σας ερωτώ, Ο ΟΠΕΚ τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό. Επίσης, τελευταία ερώτηση. Πρέπει να έχουμε περισσότερε ενώσιμε πηγέ ενέργεια στην Ευρώπη, αλλά επίση θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πάντα ενεργειακό πόρο που βρίσκεται στην ε, διάθεσή μα και τα ανανεώσιμα και όλα. Επομένω, το μήνυμα των όσων μας είπατε είναι ότι θα πρέπει να μην αποκλείσουμε οποιαδήποτε πω, να μην βιαστούμε τέλο πάντων να αποκλείσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα που έχουμε. Ένα δίλεπτο κύριο Τούρμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζομαι τόσο πολύ. Λιγότερο θα χρησιμοποιήσω και θα αντισταθμίσω το ότι τα παρα, το παράκανα πριν. Σα ευχαριστώ για όσα μα είπατε όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, όσον αφορά το πετρέλαιο και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν μπορείτε να, να μας τα ξαναεξηγήσετε δηλαδή γιατί αυτές οι νέες τεχνολογίες χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την παραγωγή της Αυγής Αραβίας για πέστε μας για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο τι γίνεται με την ε, Αμερική εγώ νομίζω ότι πρόκειται εκεί πέρα για κάποια φούσκα και όχι οτιδήποτε άλλο γιατί η συμβατική παραγωγή, το συμβατικό αέριο εκεί παράγεται όλο ένα και λιγότερο. Και εσείς πώς τα, πώς τα βλέπετε τα θέματα. Αν έχουμε μένω την, ε, την παραγωγή όπως και στο θα αυξηθεί η παραγωγή. Τι θεωρείτε ότι θα γίνει στη ΣΥΠΑ όταν ε, σκάσει, σπάσει τέλο πάντων αυτή η φούσκα της παραγωγής του αερίου. Λάμστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας είπατε μας ότι σε 60 χώρες μειώνεται η παραγωγή. Σε 60 χώρες όλο τον κόσμο. Έχουμε κάποιες δυσκολίες με την ε, παράδοση τέλο πάντων του φυσικού αερίου. Και επ' αυτού έχω δύο ερωτήσεις. Υπάρχει θέμα περιβαλλοντικό με την ε, άντληση με το πετρελαίου του 25% των αποθεμάτων τώρα βρίσκονται ε, στην περιοχή της Αρκτικής. Οπότε από εκεί θα ξεπηγάσουν διάφορα προβλήματα για το περιβάλλον εάν πάμε να αντιλήσουμε πετρέλαιο, να εξορίξουμε πετρέλαιο στην Αρκτική. Τι γίνεται με το μεθάνιο. Υπάρχει μια προβληματική γιατί έχει αποδειχθεί ότι έχουν γίνει κάποιες έρευνες στην Ρωσία ότι υπάρχουν αποθέματα μεθανία που λένε ότι μας αρκούν για 400 χρόνια. Αλλά και εδώ έχουμε προβλήματα για το περιβάλλον. Γιατί αυτά τα κοιτάσματα ενεργειακά θεωρούνται πλούσια και βρίσκονται στην περιοχή αυτή του Περμαφρόστ, αυτής της μονίμως, του μονίμως παγωμένου εδάφους. και έχω απευθυνθεί σε διάφορες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θεωρούν ότι τώρα είναι αντικείμενο ενδιαφέροντος ε, εκμετάλλευση κλπ. Εσείς ως ειδικό, μήπως μπορείτε να μας πείτε. Έχετε κάνει κανέναν υπολογισμό, κάποιες α, ε, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτά τα κοιτάσματα από θέματα μεθανίου. Κυρία Κάπελ, κύριε καθηγητά, ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε για το φάσμα των τιμών εντός του οποίου μπορεί να είναι αποδοτική η παραγωγή, δηλαδή μεταξύ 77 και 120 δολαρίων. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε πως η μεγάλη στρατηγική στο πλαίσιο της ε, ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να είναι η διαφοροποίηση και εδώ πέρα βεβαίως μιλάμε πάρα πολύ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ζήτημα λοιπόν είναι πως η παραγωγή αυτή επιδοτείται πάρα πολύ γιατί δεν είναι δυνατόν να καλύψει ε, το κόστος της. Το ερώτημά μου είναι τι μπορούμε να κάνουμε, πως κατά την άποψή σας θα ήταν αναγκαίο να γίνουν κάποια βήματα έτσι ώστε η διαφοροποίηση αυτή να είναι μόνιμη και βιώσιμη. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε την δυνατότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να επιβιώσουν στην αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν συμφωνώ με τον ομιλητή. Εάν οι τιμές του φυσικού αερίου πέσουν, τότε ε, τα διηληστήρια θα χρεοκοπήσουν, κάποια άλλα θα πάρουν τη θέση τους, αγορά λέγεται. Και δεύτερον, αν κάποιος είναι κατά του σχιστολιθικού αερίου, του άνθρακα και της πυρηνικής ενέργειας, είναι είτε ηλίθιος είτε πράκτορας της Gazprom. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ε, Κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είπατε πως τόσο υψηλό, όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο το καλύτερο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, βλέπουμε ότι έχουμε και κάποιες εμπειρίες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους μας. Οπωσδήποτε υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες στρεβλώσεις, υπάρχουν κάποια κράτη όπου η τιμή των ορυκτών καυσίμων είναι τόσο χαμηλή που αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και αυτό μπορεί να οδηγήσει ε, στο ότι δεν θα ξέρουμε για τι θα γίνει για αρκετά χρόνια, να οδηγηθούμε σε στρεβλώσεις της αγοράς και βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ πέρα η στήριξη των ανανεώσιμων. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Δεν βλέπω. Ωραία. Να ζητήσω τις απαντήσεις παρακαλώ. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω τις δικές μου ταπεινές ε, συνεισφορές και απαντήσεις σε αυτά που τέθησα. Πρώτα απ' όλα για την ε, πολιτική πίεση. Είπαμε, ποιες είναι οι τάσεις, οι οποίες είναι πολύ κειμενόμενες βέβαια και μεταβλητές μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, αλλά υπάρχουν πολλές υποθέσεις και στοιχήματα για το τι θα γίνει από πολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή παντού λέγεται ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να χειριστεί την αγορά για να πλήξει τους Ρώσους ή την, τον ανταγωνισμό, να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από το πετρέλαιο το σχιστολιθικό των Πολιτειών. Πιθανόν, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν προσπάθειες να χειριστεί κανείς την αγορά αλλά πρέπει να είμαι κανείς πολύ προσεκτικός γιατί γι' αυτό δεν έχουμε πληροφορίες. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε και μπορούμε να μετρήσουμε είναι το κόστος της παραγωγής. Αυτό αυξάνεται και αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Εάν μου επιτρέπετε, σκεφτείτε, είναι σαν να οδηγεί κανείς ε, κάποιο, να οδηγεί Φόρμουλα 1. Μπορεί να είναι φοβερός οδηγός, αλλά αν δεν είναι αρκετά γρήγορο το αμάξι, δεν κερδίζει κανείς Εδώ ε, βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί κανείς να προσπαθήσει να χειριστεί την αγορά, αλλά πόσο. Λίγο ναι, πολύ όχι. Αυτός ο μύθος για τη Σαουδική Αραβία ε, δεν μπορεί να ισχύει απολύτως, διότι αν η Σαουδική Αραβία θέλει μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της. Δείτε εσωτερικώς τι συμβαίνει και εκεί υπάρχουν δυσκολίες το πετρέλαιο είναι ακόμη φτηνότερο από ότι το ρωσικό, που είναι πολύ φτηνότερο από το αμερικανικό. Αλλά το πρόβλημα είναι ακριβώς και αυτή η εξάντληση των κοιτασμάτων που είπαμε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί κανείς να αυξήσει όσο θέλει. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά σήμερα εκτιμάται ότι έτσι παρουσιάζουν τα κοιτάσματα πετρελαίου τους. Ναι, σωστό και αυτό. Οι πληροφορίες που έχουμε στην πραγματικότητα από χώρες της Μέσης Ανατολής είναι λίγο αποσπασματικές. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια ερμηνευτική για να καταλάβει κανείς τι γίνεται εκεί. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι κοντά στα όρια τους. Οι Σαουδαράβες δεν μπορούν να αυξήσουν πολύ περισσότερο από αυτό που παράγουν τώρα. Σε κάθε περίπτωση η δική μου οπτική κοιτάζει περισσότερο το μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα όλοι θα έχουν πρόβλημα να αυξήσουν την παραγωγή του. Σε μια άλλη ερώτηση για τι ανανεώσιμε πηγέ. Εάν οι ανανεώσιμε πηγέ μπορεί να είναι ανταγωνιστικέ ω προ τα καύσιμα. Ε, Καλή ερώτηση, γιατί έχει εξελιχθεί και έχει βασιστεί όλη μα η κοινωνία στα ορεικτά καύσιμα εκεί βρίσκονται τα θεμελιά μας και όλο μας το οικοδόμημα. Αν δούμε όμως το γνωστό ε, δίκτυ ή ρόη όπως λέγεται, την καθαρή απόδοση της ενέργειας, θα δείτε ότι οι ανανεώσιμες ε, δίνουν ε, περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα από τα ορυκτά καύσιμα, όμως δεν έχουμε τις υποδομές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τις εντάξουμε. Ε, και να έχουμε μια καλή συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στο energy mix που θέλουμε. Οι μεταφορέ μα ε, κατά κύριο λόγο βασίζονται στο ρηκτά καύσιμα, στην, ε, στο πετρέλαιο, τη βενζίνη δηλαδή. Εάν προσπαθήσουμε να περάσουμε από τα φορτηγά στους σιδηροδρόμους, από τα αυτοκίνητα, στα ηλεκτροκίνητα τρένα, είναι τεράστια η επένδυση και σας καλώ να το σκεφτείτε. Ποιες θα ήταν οι εναλλακτικέ μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την εξάντληση των κοιτασμάτων. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε την πολιτική μας βούληση για να μην υπάρξει εξάντληση κοιτασμάτων, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς ιδεολογικά κολλήματα. Είναι ένα πρόβλημα που είναι επαρκτό. Θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε βασικές δυνατότητες, ένα δυναμικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε σε μελλοντικές κρίσεις. Ήδη είχαμε αρκετή κρίση φέτος. Και σίγουρα θα έχουμε και περισσότερα προβλήματα στο μέλλον. Οπότε ένα βασικό στοιχείο της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη είναι να έχουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να παράγουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη. τέτοιες δυνατότητες μεγάλας, μεγάλα εργοστάσια υπάρχουν στην Νότια Αφρική λόγου χάρη για την ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορούσε να εξαγεται στην Ευρώπη. Βέβαια αυτό σημαίνει πια άλλη μια σχέση εξάρτησης. Αλλά έγινε και μια πολύ καλή παρατήρηση, δηλαδή εάν οι τιμές του πετρελαίου πέσουν, σημαίνει αυτό ότι ίσως ο ανταγωνισμός των ανανεώσιμων τελικά πετυχάνει το στόχο του. Όχι όμως, γιατί πέρα από τα παραδοσιακά, ε, ε, τις παραδοσιακές ανανεώσιμες, όπως η υδροηλεκτρική, <clears throat> οι υπόλοιπε, ηλιακή και αιωλική, είναι ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι ότι η ζήτηση μειώνεται. Εάν δείτε τι γίνεται στην Ιταλία, χώρα που γνωρίζω καλά, η ζήτηση πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 35% τα τελευταία χρόνια. Καταναλώνουμε λιγότερο. Όλοι οι Μεσόγειος, οι μεσογειακές χώρες της Ευρώπης γνωρίζουν κατάρρευση στην αγορά τους λόγω της μείωσης ε, της κατανάλωσης ενέργειας φοβερό περιορισμό τη ζήτηση. Γι' αυτό πέφτουν και οι τιμέ του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπαραγωγή πετρελαίου σε σχέση με το ότι μπορεί να καταφέρει να αγοράσει κανεί στην αγορά με τι τιμέ γύρω στα 100 πριν από λίγου μήνε. Λίγο παραπάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Χώρες όπως η Ιταλία δεν μπορούσαν να το καλύψουν το κόστος. Έγινε και άλλη μια παρατήρηση, γιατί αυτές οι νέες τεχνολογίες καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Καλή ερώτηση, διότι η τεχνολογία της εδρορογμάτωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκη, είναι φανταστική, είναι υπέροχη κατά μία έννοια, διότι δεν κάνει κανείς μια τρύπα απλώς στο έδαφος, αρχίζει μια κάθετη εξόριξη και ξαφνικά αυτή γίνεται οριζόντια και προσπαθεί με ένα τρυπάνι, ε, με ένα black σαν black and decker να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο το πρώτο σημείο εισόδου, διότι αν αντλήσει κανείς με υψηλή πίεση και βάλει ε, με δύναμη τα, το υγρό που χρειάζεται για να σπάσει το πέτρωμα, δεν πετυχαίνει. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν. Είναι φανταστικό αυτό που κάνουν. Αλλά είναι ακριβό, μπορείτε να το φανταστείτε. Το γεγονός ότι το αέριο ο σωστός όρος δεν είναι το shale gas, είναι tight gas το σχιστολιθικό αέριο. Είναι πολύ φτηνό στις ΗΠΑ το αέριο αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπαραγωγή και όποιος ορθώς είπε κάποιος πρόκειται για χρηματοοικονομική φούσκα, ε, διότι η βιομηχανία απορροφά τις επενδύσεις προς τη ε, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, προσδοκώντας ότι θα έρθουν ε, πολύ καλές στιγμές στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο και το αέριο αυτό δεν αποθηκεύεται. Πρέπει να πουληθεί και πωλείται σε χαμηλή τιμή. Πρόκειται όντω για φούσκα, διότι είναι πολύ εμπορευόμενοι που πουλάνε με ζημιά. Αυτό συνεχίζεται λόγω των οικονομικών συνθήκων. Όμως, ναι, ναι, ναι, θα οδεύσω προς τα συμπεράσματά μου. Όταν θα σκάσει αυτή η φούσκα και πότε, πολύ ωραία ερώτηση, αν ξέρει κανείς θα ήθελα και εγώ την απάντηση. Πολλά, πολλά ακόμη. Ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο για το αέριο από μεθάνιο. Νομίζω ότι είναι υπερεκτιμημένα αυτά τα κοιτάσματα. Υπήρχαν πάρα πολύ υψηλές εκτιμήσεις για αυτό το μεθάνιο στις περιοχές με μόνιμους παγετώνες θα ήταν καταστροφική όμως η αξιοποίησή του για τους, ε, από την σκοπιά της επερθέρμανσης του πλανήτη και των κλιματικών αλλαγών. Αυτού του είδους οι εκμεταλλεύσεις θα κατέστρεφαν ένα σωρό περιβαλλοντικά στοιχεία. Και ε, τελευταία ερώτηση, πώς, μπορεί να γίνει μπορούν να, να γίνουν ανανεώσιμες ανταγωνιστικές. Μα να σταματήσουν οι επιδοτήσεις. Είναι νομίζω η καλύτερη λύση. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε ε, μήπως κάποιες επιδοτήσεις πρέπει να παραμείνουν. Η χρηματοοικονομική αγορά πρέπει να πιστέψει και να επενδύσει στην αγορά αυτή. Ε, είναι κερδοφόρα αγορά η επιλογή για επενδύσεις μεταξύ πετρελαίου ή ανανεώσιμων είναι μια επιλογή που την κάνει η αγορά. Θα πρέπει να είμαστε ευφύ και να οδεύσουμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Διότι μπορεί κανείς να κερδίσει πολλά με τις ανανεώσιμες. Αλλά έχω και μια απάντηση για τον κύριο είπε ότι διαφωνεί μαζί μου, αλλά η ερώτησή σας χάθηκε στην μετάφραση, οπότε αν θέλετε να το συζητήσουμε διμερώς μετά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εξαιρετικές ε, ομιλίες, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λέγονται, δύσκολο να σας διακόπτω ε, επειδή είσαστε και οι βασικοί ομιλητές. Σας ευχαριστώ και τους τρεις, διότι τώρα η σύνθεση του πάνελ θα αλλάξει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κυρία Σβέντας, κυρία Μπράτουσκα και κύριε Μπάρντι. Σας ευχαριστούμε για τις ομιλίες σας, για τις απαντήσεις σας και τώρα θα ζητήσω από την κυρία Φουκέ και τον κύριο Ρίνας και τον κύριο Έλενας να έρθουν για τις παρουσιάσεις τους. Να περάσουμε από το θέμα του πετρελαίου στο αέριο. CEO για τους υδρογονάνθρακες. Ε, παρουσίαση του κυρίου Ελλήνας για τις ε, ενεργειακές πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο και τον εντατικό διάλογο με τους εταίρους μας της Ανατολικής Μεσογείου με σκοπό τη δημιουργία ενός κόμβου για το αέριο στη Μεσόγειο. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το θέμα σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι ευχαριστή για μένα να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα να σας μιλήσω για αυτό το ζήτημα το οποίο νομίζω μπορεί να συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Τα θέματα τα οποία θα ήθελα να καλύψω σήμερα είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε για τις ενεργειακές πηγές στην ε, Ανατολική Μεσογείο. Υπάρχουν ε, αρκετέ πηγέ αερίου και φυσικού αερίου που, αν αναπτυχθούν σωστά, μπορούν να συνεισφέρουν στην ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ το 2010 υπολόγισε πω η λεκάνη του Λεβάντε έχει μέσα πιθανά πετρελαιακά αποθέματα 1,7 δισεκατομμυρίων βαρελιών και μη ανακαλυφθέντα ακόμα αποθέματα φυσικού αερίου 3,5-3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Οπότε ε, υπολόγισε ακόμα πως ε, τα μέσα μη ανακαλυφθέντα ακόμα αποθέματα υγρού φυσικού αερίου είναι στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν όλα αυτά έρθουν στην Ευρώπη, μιλάμε για 20% των τρεχουσών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φυσικό αέριο. Με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μισές από αυτές τις πηγές ενέργειας είναι ευρωπαϊκές. Μέχρι τώρα, με κάποιες ερευνητικές γεωτρήσεις που έχουν γίνει στην Ισραηλινή και την ε, Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη που είναι το 1 τρίτο της λεκάνης Λιωδάντα έχουμε φτάσει γύρω στα 1200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου οπότε είναι από ό,τι φαίνεται αρκετά α, μεγάλα τα κοιτάσματα εκεί πέρα με 1.700 δισεκατομμύρια βαρέλια στην Κύπρο, ανάλογες ποσότητες στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Και ακόμα Έχουμε το Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο που υπολογίζεται ότι περιέχει ακόμα μεγαλύτερε ποσότητε. Οπότε και τα έξι μπλοκ τα οποία αυτή τη στιγμή έχει μισθώσει η Κύπρο στην ΑΟΣ πιθανώ να περιέχουν ε, χίλια δισεκατομμύρια βαρελιά. κυβικού. Ε, με χίλια ε, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα κυβικού αερίου. Οπότε βλέπουμε ακριβώς την ΑΟΣ της ε, Κύπρου και την λεγόμενη λεκάνη του Λεβάντε. Τα έξι μπλοκ τα οποία έχουμε μισθώσει είναι το υπαριθμόν 12, το οποίο εκμεταλλεύεται η Νόμπλα Τσίπα. Και μετά έχουμε τα οικόπεδα 2, 3, 5, 9 και 11, τα οποία εκμεταλλεύονται ευρωπαϊκές εταιρείε, η ΕΝΗ και η Total. Η ανακάλυψη των αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένας καταλήτης ευρύτερης συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο που θα συνεισφέρει βεβαίως στην ειρήνη και σταθερότητα την περιοχή. Γνωρίζετε βεβαίω τα προβλήματα με την Τουρκία που επηρεάζουν την κατάσταση. Η Τουρκία δεν έχει προβλήματα μόνο με την Κύπρο και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ έχει προβλήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει κάποια περιφερειακή συνεργασία για την ενέργεια και εντατικοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της Μεσογείου απέναντι στην ρήπανση που προκύπτει από τέτοιες δραστηριότητες. Η ανάπτυξη αυτών των πόρων θα πρέπει να είναι για το όφελος της Κύπρου και ελπίζουμε να αποτελέσει κίνητρο για την επίλυση του Κυπριακού έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφεληθούν όλοι οι Κύπροι. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι εταιρείε Noble και και δεδομένη της προχωρημένη φύση των ερευνών τους στο Ισραήλ και στην Κύπρο και το τι θα κάνουν θα επηρεάσει τι μελλοντικέ εξελίξεις. Οι Ένι με την Κόγκα ακολουθούν μετά καθώς έχουν ένα πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων στα οικόπεδα 2, 3 και 9, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο εξάμεινο 2016. Η Total σκοπεύει να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμεινο 2015. Η Αίγυπτος πρόσφατα δημοπράτησε νέα οικόπεδα υπεράκτια και τα πήραν και η ΕΝΗ και η Total μεταξύ άλλων. Επίση, σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων έχει οδηγήσει σε αναζωπήρωση παραγωγή φυσικού αερίου και το Λίβανο ακολουθεί κατά πόδας αλλά ακόμα απέχει. Στο Ισραήλ, ε, το Ισραήλ είχε αυτό το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρήσα, θεωρήσαμε το μεγαλύτερο υπεράκτιο πεδίο φυσικού αερίου. 500 δισεκατομμύρια δηλαδή κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η φάση 1 έχει ήδη ανακοινωθεί και θα βασιστεί σε ένα σχήμα το οποίο θα παράγει γύρω στα 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο για τη Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ορδανία και Αιγυπτό στα σχετικά τους ε, σχετικές εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η επόμενη φάση είναι του χρόνου και θα μπορούσε να οδηγήσει εξαγωγές στην Τουρκία μέσω Κύπρου για τα επόμενα 30 χρόνια και αν δεν ε, επιτύχει αυτό ίσως πάνε σε κάποιες άλλες ε, επιλογές. Στην Αίγυπτο τώρα. Η, Αίγυπτο, μιλάμε, η Αίγυπτος μιλάμε ότι έχει γύρω στα 2.200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποδεδειγμένα κοιτάσματα, όμως αυτή τη στιγμή τελευταία χρόνια βεβαίως φαντάζεστε το επενδυτικό περιβάλλον δεν είναι το καλύτερο και έχουμε οδηγηθεί σε μια στασιμότητα, κάτι το οποίο βεβαίως θα αλλάξει δεν Υπάρχει μια αναζωπήρωση της δραστηριότητας και τα επόμενα πέντε χρόνια η Αίγυπτος θα φτάσει να εισάγει αέριο και αυτή τη στιγμή αγοράζουν LNG από την Αλγερία αλλά και από το Ισραήλ, από την Ταμάρ. Οι δυνατότητες ε, των ε, δύο εγκαταστάσεων LNG της Αιγύπτου είναι γύρω στα 12 εκατομμύρια ε, τόνους ε, ε, και αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούν γύρω στο 25% της δυναμικότητάς τους μια Βρετανική και μια Ισραηλινή εταιρεία. Εάν ξεκινήσει λοιπόν η πλήρης εκμεταλλευσή τους θα μπορέσουν να επαναλάβουν τις εξαγωγές τους και στην Ευρώπη. Στην Κύπρο η Νόμπλ εξετάζει λεπτομερώς όλες τις πιθανές εξαγωγές από το πεδίο της Αφροδίτης στο οικόπεδο 12 και παρουσίασαν τα αρχικά τους ευρήματα στην κυβέρνηση της Κύπρου τον Οκτώβριο. Λόγω των ποσοτήτων προτιμάει η Νόμπλ να κάνει εξαγωγή στην περιφερειακή αγορά, στη Μεσόγειο, είτε μέσω CNG, είτε μέσω αγωγών. Μάλιστα θα προτιμούσαν να, το αγοράσει κάποιος από τις εγκαταστάσεις τους και να αναλάβει, να αναλάβει ο πελάτης την ευθύνη της παράδοσης. Τώρα για τις ε, χερσαίες εγκαταστάσεις ε, LNG στην Κύπρο είναι κάτι το οποίο θα επανεξετάσουμε μόλις ξεκινήσει η άντληση. Η Κύπρος βεβαίως ως κάρτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πολύτιμο αγωγό για την ροή φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσογείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο διάδρομος της Ανατολικής Μεσογείου θα οδηγούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Είχαμε κάποια έργα το 2012, αλλά αυτά τα οποία προτείνονται δεν είναι πάρα πολύ πρακτικά. Δηλαδή μιλάμε για έναν αγωγό από την Κύπρο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αφενός ε, είναι στη θάλασσα, μεγάλο το κόστος, τεχνολογική δυσκολία. Βεβαίω ο μεγαλύτερος όγκος ακόμα δεν έχει ε, αποδειχθεί ότι υπάρχει και θα είναι στα υπόλοιπα πέντε οικόπεδα της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ. Έχουμε ακόμα ερευνητικές γεωτρήσεις και θα επιβεβαιώσουμε τις ποσότητες ε, μέχρι το 2018-2019. Οι επιλογές μας μάλλον θα είναι προς το LNG το υγροποιημένο φυσικό αέριο και είτε θα έχουμε χερσαίες εγκαταστάσεις είτε πλωτές. Η ευελιξία του LNG βεβαίως μπορεί να διευκολύνει τις απαραίτητες επενδύσεις για την εφαρμογή του διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου που θα καταστήσει την Κύπρο κόμβο για την περιοχή. Έτσι θα μπορούσε να μεταφερθεί το αέριο στην Νότια Ευρώπη. Συμβολή τώρα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η κρίση της Ρωσίας και Ουκρανίας ε, έχει φέρει στο προσκήνιο την... Ε, το πόσο η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ευάλωτη καθώς δεν είναι συνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το αέριο λοιπόν από το πεδίο της Αφροδίτης μπορεί να βοηθήσει αυτές τις χώρες ήδη από το 2018. Δεδομένων των υφιστάμενων αποθεμάτων θα μπορούσαμε να μιλάμε για 7 ως 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο και άρα τα κράτη-μέλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα μπορούσαν να έχουν ενεργειακή ασφάλεια που δεν προσέφερε ο Ναμπούκο και σε λίγα χρόνια να κάνουμε και εξαγωγές. Όπως βλέπετε από τον πίνακα αυτών. μιλάμε για το μισό φυσικό αέριο που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή οι χώρες αυτές από τη Ρωσία. οι μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές όσον αφορά την τιμή του υγροποιημένου φυσικού που θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της δεκαετίας και πιθανώς και παραπέρα πέφτουν οι τιμές του αερίου και σε μορφή LNG και είχαμε μακροπρόθεσμες αλλαγές ε, στις ασιατικές αγορές λόγω της ουκρανικής κρίσης. Οπότε η αυξανόμενη συνεργασία Ρωσίας με την Κίνα και η στροφή της Ρωσίας στην Ασία είναι μόνιμη, κάτι το οποίο έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η Κίνα πλέον γίνεται μακράν η πιο κυρίαρχη αγορά ενέργειας ε, και μια που έχουν υπογράψει με τους Ρώσους ή παγορεύουν τι τιμέ. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή υπερβολική προσφορά LG σπαγόσμε αγορέ. Οπότε η υπαγορεύουν τις τιμές. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή υπερβολική προσφορά LNG στις παγκόσμιες αγορές, ε, οπότε η τιμή πρέπει να είναι σωστή. Κανείς δεν αγοράζει σε οποιαδήποτε τιμή, δεν είναι θέμα πολιτικής ε, βούλησης, πρέπει να υπάρχει μια εμπορική τιμή. Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξελίξεις γρήγορα. Μπορεί τα περσινά μας σχέδια πλέον να μην ισχύουν πια. Ένα λεπτό ακόμα έχει το λέει, ο πρόεδρος. Λοιπόν, κοιτώντας το μέλλον, το σαφές είναι πως ε, η παγκόσμια αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου υφίσταται ταχύτατες αλλαγές. Ε, τα καλά νέα είναι πως μόλις ξαναξεκίνησαν οι γεωτροί στην Κύπρο, στην ΑΟΣ. Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει με το να στηρίξει την συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, Λιβάνου και Ελλάδας και να βοηθήσει την επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία και η Κύπρος θα υποφεληθεί από μακροπρόθεσμα σχέδια και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για να, επενδύσει, για να προσελκύσει επενδύσεις. Τέλος, τελευταία σελίδα μάλιστα, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο οικόπεδο 12 μέσω περιφερειακών εξαγωγών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και μετά μπορούμε μέχρι το 2018 να ξεκινήσουμε εξαγωγές συνεισφέροντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Οι επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων νομίζω θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας και επίσημη αναγνώριση του διαδρόμου αυτού από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενέργειας νομίζω θα αποδώσουν στο θέμα αυτό τη σημασία που το αξίζει. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα ο εισηγητή μα θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Σαουδάργας, σας ευχαριστώ για την εισηγησή σας. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα που σας αφορά. στον τομέα που μας αναλύσατε, γιατί βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες, όσον αφορά το ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ ε, ε, λύσεις και, και για τους ενδιακούς πόρους και διαφορετικοί πόροι. Γιατί η Κύπρος έχει σημαντική θέση, αλλά τέλος πάντων μας αναφέρατε το Ναμπούκο και το θέμα του νοτίου διαδρόμου ε, το South Stream επίσης και πάλι εδώ μπαίνει το θέμα του ρόλου της Ρωσίας ε, αναφέρετε και κατονομάσατε χώρες την Τουρκία, το Ισραήλ την Αίγυπτο και σας ρωτώ εσείς πώς το βλέπετε τι θα πρέπει να κάνουμε τόσο ώστε να έχουμε κάποιο είδους πολιτική σταθερότητα Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να πει ότι όλα αυτά είναι συνταγή για πολιτική αστάθεια. Εσείς τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το αντίθετο. Thank Mr. Chair. I have a very short question. How do you evaluate the potential... Δεν μου λέτε. Δεν υπάρχει εδώ ένας ενδεχόμενος κίνδυνος. Δηλαδή το να πρέπει να έχουμε κάποια τεράστια υπερπαραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε τον τερματικό για το υγροποιημένο αέριο και πάμε για τα 25-27% που θα περάσουν από εκεί. Ήδη έχουμε επομένω ε, υπερπαραγωγή όσον αφορά την προσφορά. Μα γιατί να έχουμε τόσο μεγάλες επενδύσεις ενώ ήδη υπάρχει τόση υποδομή, γιατί να πρέπει ο, Ευρωπαίος να πληρώσει για τέτοιου είδου ε, επενδύσεις. Κύριε Σιλικιώτη, Σιλικιώτη έχετε λόγο. Ε, το ερώτημα προς τον κύριο Έλληνα είναι ε, τι θα αναμένει κάποιος για, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη στήριξη για τις υποδομές. γνωρίζουμε πολύ καλά ότι Υπάρχει το πρόγραμμα Συνδέοντας στην Ευρώπη, υπάρχουν προτάσεις κατατεθειμένες και ε, πώς πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να στηρίξει υποδομές στην περιοχή οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια. Και το δεύτερο ερώτημα είναι σε σχέση με την συνεργασία με τις χώρες της περιοχής. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, και το Ισραήλ ε, και η Αίγυπτος αναμένεται στο μέλλον ενδεχομένω ο Λίβανο να εξεύρουν σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Ε, πώς πρέπει, μέσα από ποιε διαδικασίε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει συνεργασία με τι χώρε τη περιοχή ώστε να στηρίξει έτσι την ενεργειακή ασφάλεια τη Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε το Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα κύριε Έλληνα, με εντυπωσίασε η εικόνα που δώσατε για τις μέλους ε, εξελίξεις και σας ερωτώ με τέτοιες εξελίξεις μπορούμε να ελπίσουμε σε ε, μια διέξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση, δηλαδή με τέτοιους ε, ενεργειακά αποθέματα. Άλλη παρατήρηση. Αναφέρατε το Ισραήλ. Μήπως θα πρέπει να διορίσουμε αυτό το οποίο λέγεται για την Golda Meir που είχε πει, λένε κάποτε, ότι ο Μωυσής ήταν ηλίθιος γιατί πήγε τους ε, Ιουδαίους τότε στην μόνη χώρα της Αγγής Ανατολής όπου δεν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Ε, Mr. Fox. Fox. Thank you, President. Και εσείς είστε σχεδόν εισηγητές μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Φόξ, ευχαριστώ για την εισήγηση, κύριε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πεπερασμένα χρήματα, πεπερασμένους πόρους για να μπορέσει να βελτιώσει την ενεργειακή υποδομή ε, και να έχει διασυνδέσεις στους αγωγούς. Προτεραιότητά μου θα ήταν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για να βελτιώσουμε την ενεργειακή ασφάλεια στην ε, ε, ένωση και να έχουμε μια ενιαία αγορά στην ενέργεια ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα εμπόριο εσωτερικό μεταξύ μας. Εσείς, ποια έργα ή προγράμματα θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να πετύχουν αυτό το στόχο. Μήπως αντικειμενικά δικαιολογείται η χρήση των ε, ενωσιακών πόρων για τους αγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρείτε ότι είναι πιο εύστοχη αυτή η επένδυση από το να έχουμε κάποιο είδου διασυνδεσιμότητα μέσα στην Ευρώπη τώρα. Any other requests? Ζητεί άλλο το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Ιαννή. Όχι από ό,τι φαίνεται. Κύριε Έλληνα, αν θέλετε απαντήστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πω ότι είναι μια χώρα στην περιοχή που συνεργάζεται στενά με την Κύπρο. Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανο. Εδώ υπάρχει ένας βαθμός συνεργασίας με κέντρο της συνεργασίας αυτής στην Κύπρο. Η μόνη χώρα που αρνείται στεναρά να συμμετάσχει είναι η Τουρκία, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με την Κύπρο. Η Τουρκία έχει τα ενεργειακά μέτρα σαν τα δικά τη. και εάν δεν λυθεί το Κυπριακό είναι πολύ δύσκολο να γίνει οτιδήποτε. Με, τα, με τις ανακοινώσεις που έχουν ε, γίνει για το χρόνο θα μπορούσαν να υπάρξουν σοβαρέ ε, πωλήσει αερίου προ την Τουρκία αρκεί να λυνόταν το Κυπριακό. Υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες να λυθεί εδώ το θέμα ε, όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλλά αν ο δρόμος για τις εξαγωγές αερίου από το Ισραήλ στο, στην Τουρκία ανοίξει τελικά και εφόσον κλείσουν κάποιες πολιτικές προποθέσει, θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η λύση. Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σταθμούς που λαμβάνουν το LNG, το ευρωποιημένο φυσικό αέριο, θα μπορούσε να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες αρκεί να φτάνει κάποτε και το υγροποιημένο φυσικό αέριο από κάπου στους σταθμούς αυτούς, στις εγκαταστάσεις, από την Αίγυπτο και την Κύπρο λόγω χαρά την Ανατολική Μεσόγειο. Ως προς την ε, ενίσχυση της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις επενδύσεις που χρειάζονται ε, με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τεράστιες οι επενδύσεις αυτές. Εάν αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες της περιοχή και συμβάλλει κανεί στην επίλυσή τους, χρειάζεται και κάποια οικονομική στήριξη που θα βοηθούσε αλλά όπως έχω πει και προηγουμένως, ε, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υπάρχει ένας αποκλεισμό. Δεν επωφελείται η Νοτιοανατολική Ευρώπη από το αέριο που φτάνει στην Δυτική. Ε, εξαρτώμεθα από το ρωσικό αέριο και δεν υπάρχουν και πολλέ επιλογέ. Ήδη τον τελευταίο μήνα η Βουλγαρία έφτασε στο Αζερμπαϊτζάν για να εξασφαλίσει ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα αερίου ε, είναι αστείο. Είναι πολύ ε, μικρό το ποσό και χρειάστηκε να πάει στην Πακού για να το εξασφαλίσει από τον αγωγό που είναι πρόσφατος. Ε, θέλουμε λοιπόν αέριο ανεξαρτήτως και από τη Ρωσία, όχι αναγκαστικά για να μην έχουμε καμία σχέση με τη Ρωσία, αλλά για την αυταρκιά μας. Η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος είναι σε πολύ καλή θέση για να παράσχουν αυτό το αέριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα η Ευρώπη θα μπορούσε να υποφεληθεί στηρίζοντας αυτές τις εξαγωγές αερίου προς την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη ώστε να ε, οδεύσουμε προς την Ενεργειακή Ένωση και την Ενεργειακή Ασφάλεια. Για να ολοκληρώσω λοιπόν τη στιγμή που αναζητά την Ενεργειακή Ασφάλεια και φτάρει και η Ευρώπη, είναι σημαντικό η Ανατολική Μεσόγειος και ο διάδρομός της να μπουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Αγορά οι ποσότητες αερίου που υπάρχουν είναι σημαντικές και μπορούν να ε, συμβάλλουν στην ασφάλεια των χωρών στην νότια-ανατολική και νότια Ευρώπη. Εκεί που υπάρχει λιγότερη ευελιξία για την πρόσβαση στο ρωσικό αέριο. Ε, το αέριο αυτό είναι ευρωπαϊκό στην πραγματικότητα. Τα κοιτάσματα αυτά είναι ευρωπαϊκά. Ε, Όπω είπα κάποιο σήμερα νωρίτερα, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλου του διαθέσιμου πόρου. Ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγουμένως, πρωτού στραφούμε προς τα έξω. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές του αερίου πέφτουν. Η διαφορά των τιμών Ευρώπης-Ασίας είναι πολύ μικρότερη από ό,τι πριν από λίγα χρόνια το να ε, αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό αλλά για την ώρα στα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό ο διάδρομο από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ακριβώ ο διάδρομο για το σχετικό δίκτυο πρέπει να γίνει μέρο τη ε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, αλλά Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένας πρωταγωνιστής στην επίλυση των θεμάτων. Το όφελος θα ήταν η ευελτίωση της συνεργασίας, η σταθερότητα και πραγματική συμβολή στη διαφοροποίηση της ενεργειακής κατάστασης στην Νότια Ευρώπη και η επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ε, συμβολή σας και τις, ερωτα... τις απαντήσεις που μας δώσατε και για την αρχική σας παρουσίαση. Τώρα να περάσουμε στις ανανεώσιμες ε, κατά κύριο λόγο. Η κυρία Ντοέρτε Φουκέ είναι δικηγόρος στη BBH και διευθυντής της διευθύντρια μάλλον της, Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η παρουσίασή σας αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πράσινη διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στατική Ασφάλειας. Προτεραιότητα για την αποδοτικότητα, της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και τη διάσταση της ζήτησης, καθώς και τη διαχείρισή τους, μαζί με την ευφύ χρήση των διευθυντικών κονδυλίων. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Chairman, Μεγάλη μου χαρά σας μιλώ σήμερα με αυτή τη θέση κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ευγενικά τα προσεχογικά σας ε, λόγια. Έχω ενεργοποιήσει το τομέα από το τέλος δεκαετίας του 1980 να σας πω πώς βλέπουμε τα πράγματα όσον αφορά τα ανανεώσιμα και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ του στρατηγικού εγγράφου και του δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Γιατί αυτό θα έπρεπε, θα έπρεπε να είναι ένα πόσο τμήμα της πολιτικής μας για το κλίμα και την ενέργεια. Έχουμε αναλάβει κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις εδώ και πολύ καιρό και πρώτα πρώτα είπαμε ότι έχουμε υποσχεθεί σε όλο τον κόσμο ούτως ώστε να σταματήσει ε, να χρησιμοποιείται ο άνθρακας στο σύστημα μέχρι το 2050 και επίσης να ε, έχουμε αρνητικά μεγέθη εκπομπών στη συνέχεια. Αυτό όμως δεν είναι το θεματολόγιο της ε, στρατηγικής μας και του εγγράφου του σχετικού του γνωστού. Εκτός από αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το να έχουμε αυτάρικα, να έχουμε ασφαλή προσφορά και μεταφορά ε, από, την, από τις τέτοιες χώρες πέραν της Ρωσίας και οπότε θα πρέπει να σταματήσει η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει με τους αγωγούς οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτού του είδους ε, το έγγραφο ε, αφορά το θέμα της ασφάλειας και μπορεί να φαίνεται κάπως κοινικό το ότι θα πρέπει να έχουμε ε, κάποιο είδους ε, πρόγραμμα διάσωσης από πλευράς της ε, προσφοράς του φυσικού αερίου να δούμε πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να δούμε πώς ταχαίως θα εκμεταλλευτούμε, θα αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είδατε ότι έχουμε κάποιους που χρηματοδοτούνται από δικά μας χρήματα. Δηλαδή ο, η του Πούτιν είναι ένα πρόβλημα. Η λύση όμως ε, είναι το να μην είμαστε παιχνιδάκια στα χέρια του. Θα πρέπει να γίνει αποκλιμάκωση όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ της χώρας με, που έχει τέτοια προϊστορία διαφθοράς και από την άλλη μεριά έχουμε την ε, ε, αναξιοπιστία. Έτσι, έτσι έγινε με την Ουκρανία και τη Ρωσία και τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποια αποδυνάμωση της Ρωσίας από, οικονομικό, ε, από οικονομικής ε, οπτικής γωνίας. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, το ΙΕΣ θα πρέπει να έχει σαν θεματολόγιο το ότι θα πρέπει να έχουμε αύξηση της ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να μην έχουμε εκπομπές διοξιδίου όσον αφορά τα καύσιμα, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα προς μίμηση της Σουηδίας που κατάφερε να μην έχει ορυκτά καύσιμα στις μεταφορές τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι πρωτοπόρα χώρα αυτό. Χρειάζεται επίσης να έχουμε σαφείς προθεσμίες, σαφείς στόχους και χρονοδιάγραμμα, ε, να έχουμε ενδιάμεσο, ενδιάμεσο έλεγχο και ε, διαπίστωση του τι έχει γίνει και θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε την ε, ε, βαθμία κατάργηση των ορεικτών καυσίμων το 2050 όπως έχουμε δυσμευθεί να κάνουμε. Σε αυτό το έγγραφο, σε αυτή την ε, έκθεση έχουμε τους βασικούς άξονες. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το φυσικό αέριο για τα ρηκτά καύσιμα. Θα πρέπει να πάμε και ακόμα παραπέρα. Θα πρέπει να μετριαστεί η ζήτηση ενέργειας, αλλά βέβαια ε, είπαμε ότι δεν είμαστε αρκετά αυστηροί, αρκετά κατηγορηματικοί σε αυτά, δεν έχουμε ξεκαθαρό σχέδιο για την ε, αποτελεσματικότητα που θέλουμε να αποκτήσουμε. Θέλουμε επομένω μια εύρυθμη, πλήρω ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά. Ε, αυτό να καλύψει και την αγορά του ηλεκτρισμού και γενικότερα την αγορά της ενέργειας. Πάντως θα πρέπει να δούμε όλη την ενεργειακή εξίσωση την αύξηση της ενεργειακής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, σχολιάζουμε, θα πρέπει, εδώ υπάρχει κάποιο παράδοξο να σκεφτούμε. Υπάρχει κάτι το οποίο προβληματίζει, το ότι δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο ξεκάθαρη στρατηγική ουράνιο, πυρηνική ενέργεια, είναι θέματα αυτά συναρπαστικά. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Ήδη έχουμε, ξέρουμε πολλά. Αυτά που ξέρουμε όμως πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από την πορεία που χαράξαμε με τις επιτυχίες μας. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι η λύση για την ενεργειακή ασφάλεια. Κοστίζει. Πάνω από 20 χρόνια μας βαραίνει και μιλάμε για συνέπειες αρνητικές που κρατούν χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, υπάρχουν πολλές εξωτερικές πτυχές, υπάρχει, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Πάντως, τώρα η προηγούμενη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποια βήματα, έχει λάβει κάποιες αποφάσεις και τώρα έχουμε την εγγυημένη τιμή των 92,25 στερλινών ανά μεγαβατόριο. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη δεκαετία. Είπαμε για το κόστος υποδομής, πως αυτό μετακυλείται στις τιμές. Ηλιακή ενέργεια, μπορεί να δείτε εδώ τις τιμές για το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης ε, αιωλική ενέργεια για την Γερμανία. Για κοιτάξτε το γίνεται. Κάτι αποφάσισε η Γερμανία όπως και άλλες χώρες. τι αυτή η απόφαση. Όχι στα πυρηνικά, αλλά θα πρέπει να διευρυθεί το τι θα γίνει. Να βλέπετε εδώ τι γίνεται με τα ανανεώσιμα στη Γερμανία. Ανατομέα. Βέβαια δεν είναι όλα στρογγυλά και τέλεια. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για τις μεταφορές και στον τομέα της συνεργειακής αποτελεσματικότητας και στη Γερμανία. Έχουμε εδώ τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε, αλλά έχουμε και κάποιες λύσεις. Εγώ τώρα θα πάω λίγο παρακάτω. Να. Έχουμε αυτόν τον μηχανισμό στήριξης για τα χαμηλά επίπεδα, να έχουμε τις συνεργειακές πόλεις, έχουμε την σύνοδο των δημάρχων ε, από 83 ε, δήμους και κοινότητες, Φιλανδία, Βουλγαρία, Εστονία. Μιλάμε για πόλεις 8 εκατομμύριων κατοίκων. Για αυτού του είδους τα προγράμματα της βιώσιμης αηφόρου δράσης. 8 δις ευρώ. Θα απαλλαγούμε 56% από την ζήτηση του αερίου και θα έχουμε καινούργιε ε, ε, θέσεις απασχόλησης. Ως δικηγόρος βοηθώ για να έχουμε κάποιου συνεταιρισμού παντού και θα πρέπει να δούμε ότι τα ταμεία ή τόσο πάντων οι πόροι για τις υποδομές μπορούν να βοηθήσουν, είναι σημαντικός ο ρόλος τους και μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερο κεφαλαιοχικό κόστος ε, για τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. Και έτσι να έχουμε αλλαγή προς τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάποιες χώρες όπως η Πολωνία παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς έχουν χρησιμοποιήσει κάποιους πόρους για να φτάσουν στην πράσινη ενέργεια ή σε περισσότερη χρήση αυτής. Mm και άλλα προγράμματα έχουν γίνει όπως για τα δημοσία κτίρια, για τον δημοτικό φωτισμό. Υπάρχουν ε, υποτροφίες και δάνεια. Να, το παράδειγμα αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί αφορά κάποια χώρα η οποία είχε ρεκόρ χρήσης ε, άνθρακα. Ε, στην Ουγγαρία τι έγινε, έχουμε αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα όπου η θέρμανση γίνεται από βιομάζα σε ένα εντυπωσιακό ε, μέγεθος ε, δήμων και κοινοτήτων. Στην Εστονία επίσης έχουμε κάποιο είδους ε, κυκλικά αναλασσόμενο ταμείο, ε, υπόρους που προέρχονται αυτό το ταμείο. Και θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε συνολικά στο πλαίσιο της Ευρώπης και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες να δομήσουν καλύτερα, ε, να χειριστούν, να διαχειριστούν καλύτερα αυτά τα ταμεία και αυτούς τους πόρους. Ε, εδώ θα βάλω τελεία, μια που πιέζει Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ο κύριος Σαουντάργκας ως συνήθως ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την διεξοδική παρουσίαση της κατάστασης ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές. Να σημειώσω κάτι που και εσείς στήξατε, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει στη γενική μας πολιτική στρατηγική μάλλον ενεργειακή ασφαλεία, να βρούμε μια καλύτερα επικεντρωμένη στο τοπικό επίπεδο προσέγγιση. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τους υψηλά ιστάμενους, αλλά και το τοπικό επίπεδο και γι' αυτό βρίσκω εύστοχε τι παρατηρήσεις σας. Επίσης, αναφέρατε ότι υπάρχουν πολλά ισχυρά επιχειρήματα από την πλευρά των ανανεώσιμων πηγών έναντι των υπολείπων πηγών. Να αντιστρέψω όμως το επιχείρημα. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε λίγο περισσότερο την προοπτική των ανανεώσιμων. Μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές οι τιμές τους. Τι κατεύθυνση να επιδιώξουμε ώστε να υπάρξει πίστη στις ανανεώσιμες στο μέλλον και να είναι μια ανταγωνιστική πηγή ενέργειας. Ευχαριστούμε κύριο Κάριντς. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Κατάλαβα ότι ένα από τα μηνύματά σας ήταν τα πυρηνικά είναι κακά, τα ανανεώσιμα είναι καλά. Και το παράδειγμά σας ήταν η Γερμανία. Είπατε, δείτε μια χώρα που κάνει το, τη την μετάβαση στην ενέργεια πηγαίνοντας από την πυρηνική στι ανανεώσιμε. Αλλά δείτε τι συμβαίνει στην πράξη. Η Γερμανία και οι εταιρείε που παράγουν ενέργεια περνάνε από την πυρηνική στο χάλιβα. Στον άνθρακα, συγγνώμη. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το... η βασική συνέπεια των όσων συνέβησαν. Αυτό που καθορίζει τη συμπεριφορά στην αγορά είναι οι ενδείξεις ως προς τις στην αγορά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παράγουν σχιστολιθικό αέριο. Οι εταιρείε που παράγουν κλείνουν ε, τις, τα εργοστάσια που δεν παράγουν σχιστολιθικό. Οι συνολικές τιμές, ε, του, οι τιμές, του πετρελαίου παγκοσμίως πέφτουν και εμείς περνάμε περισσότερο στο χάλιβα. Αυτό συμβαίνει συνολικά. Οπότε, στον κόσμο των ανανεώσιμων, με τον οποίο δεν έχω κάποια αντίρρηση, νομίζω ότι είναι υπέροχος κόσμος, αλλά τι θα πρέπει να γίνει στον δικό μας τον κόσμο, ώστε να περάσουν οι ανανεώσιμες και εδώ και να γίνουν ανταγωνιστικές τις τιμές τους. Πώς θα γίνει μια χώρα να φύγει από την πυρηνική, να φύγει από τον άνθρακα και να παραμείνει στην αγορά ενέργειας με προσιτές τιμές από τις ανανεώσιμες. Ευχαριστούμε κύριε Λάνστορφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε ότι τα πυρηνικά εργοστάσια δεν είναι λύση για το πρόβλημα ενεργειακής ε, ασφάλειας σε εμά στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Έτσι είναι τα πράγματα, διότι στην προσπάθεια να αντιστρέψουμε τις πηγές ε, είναι πολύ ε, δύσκολο να το πετύχουμε. Έχουμε πολύ περιορισμένα κοιτάσματα άνθρακα και έχουμε αρκετά προβλήματα και με τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι καλές οι ανανεώσιμες ως συμπληρωματική πηγή ενέργειας όμως. Και θα το λέω αυτό, είναι συμπληρωματική πηγή ενέργειας, αλλά για παράδειγμα, στην περίπτωση της αιωλικής ενέργειας, τα εργοστάσια αιωλικής και ως προς την τιμή της ενέργειας που παράγουν του ηλεκτρισμού είναι 3,5%. Είναι μάλλον από 3 έως 5% ε, ακριβότερα από ό,τι συμβαίνει με την πυρηνική. Τα φωτοβολταϊκά είναι 30 φορές ακριβότερα. Ε, διότι η λειτουργία τους είναι μόνο 500 ώρες το χρόνο. Ενώ στην αιωλική 1800 ώρες το χρόνο. Η... Ε, τα στοιχεία από τη χώρα μου λοιπόν, που είναι πέμπτη χώρα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στη δική σας. Ευχαριστούμε κύριος Γιάβορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Είσαστε και η μόνη γυναίκα ομιλήτρια σήμερα το πρωί. Να έρθω σε ένα θέμα που έθιξε και προηγούμενο προκυκλημένο μα, ο κ. Μπάρντι, για το πρόβλημα των υποδομών. Είπε ότι παρόλο που οι ανανεώσιμε είναι ανταγωνιστικές και ανταγωνίζονται την πυρηνική τα ορυκτά καύσιμα, Υπάρχει το πρόβλημα των υποδομών και πώς αυτές μπορεί να αξιοποιηθούν. Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από το σύστημα των ορυκτών καυσίμων ή της πυρηνικής ενέργειας, διότι όλη η οικοδόμηση του συστήματος υποδομών μας έχει βασιστεί σε αυτές τις δύο πηγές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να έχουμε μια ενεργεια, μια σταγική ενεργικής ασφάλειας απαλλαγμένοι από την πυρηνική και τις ορεκτές πηγές. Διότι εάν εγκαταλείψουμε ε, μάλλον μήπως η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας μας οδηγεί ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Λέτε καλύτερη, περισσότερη επένδυση στις ανανεώσιμες ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά πρέπει να συνεχιστούν οι δαπάνες για τα ορυκτά καύσιμα την πυρηνική. Πώς βλέπετε να μπορεί να γίνει αυτή η εξισορρόπηση. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα που να έχει μια πολιτική διάστα, την πολιτική διάσταση της ενεργής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων και την ε, πρασινότερη πολιτική. Είναι ε, εφικτό κάτι τέτοιο ή όχι. Ευχαριστούμε κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο αφού μίλησε εδώ ο συνάδελφος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα οποία είπατε για την ανανεώσιμη ενέργεια. Καλά όλα αυτά, αλλά σύμφωνο πλήρως με τον συνάδελφο πως οι τιμές βεβαίως ε, καθορίζουν ε, και την ζήτηση και αυτό ισχύει και για εμάς στην ε, Γερμανία και αν συνέβαινε όντω αυτό με τις ε, ανανεώσιμες θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάποια ε, πράγματα γιατί δεν, όπως ξέρετε για να υπάρχει ενέργεια βάσης ε, δεν αρκούν οι ανανεώσιμες γι' αυτό έχουμε βάλει στο φουλ τα, τα εργοστάσια άνθρακα και ξέρετε τι συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού, τι έχετε να μας πείτε για αυτές τις ε, εξελίξεις και για την ε, εφοδιαστική ασφάλεια. γιατί παρόλε στις επενδύσεις, παρόλη την έρευνα δεν υπάρχει δυνατότητα ή υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα αποθήκευσης ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτι το οποίο βέβαια δεν επαρκεί ε, για να καλύψει τις ανάγκες της Γερμανίας των κατοίκων και της βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Ζωρίνιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Φουκέ για την εξαιρετική της παρουσίαση. Θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία αγορά ενέργειας που να είναι και ασφαλής και ανταγωνιστική. Αυτό είναι το θέμα κλειδί. Για να είναι και ασφαλής και ανταγωνιστική πρέπει να είναι και πολύ ευέλικτη και διαφοροποιημένη η αγορά αυτή. Όλες οι πηγές ενέργειας, όλες οι τεχνολογικές λύσεις είναι σημαντικές και πρέπει να συνδυάζονται. Σε κάθε περίπτωση τιμή των ανανεώσιμων εξαρτάται από το ευρύτερο πλαίσιο, διότι οι τιμές των ορεικτών καυσίμων επίσης εξαρτώνται από το πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να καθοριστούν οι τιμέ αυτέ. Επί πολλά χρόνια υπήρξε υπεύθυνο τη ενέργεια στην πορτογαλική κυβέρνηση και πρέπει να πω ότι ο συνδυασμό αιωλική και υδροηλεκτρική έριχνε τη μέση τιμή της ενέργειας στην Πορτογαλία. Καταφέραμε, καταφέραμε να έχουμε πολύ χαμηλές τιμές ε, στην αιωλική, 60 ευρώ το 2008 και μετά είχαμε και ένα συνδυασμένο σύστημα εκτός από τα φράγματα και αποθήκευση. Οπότε μπορούσαμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παρέχεται από την αιωλική τη στιγμή που δεν ε, χρησιμοποιείται. Όμως δεν μπορούσαμε να εξάγουμε. Οπότε ένα θέμα που πολλές φορές τίθεται είναι το κόστος των δικτύων. Άκουσα συναδέλφου να λένε ότι το 27% των ανανεώσιμων ε, σκοντάφτησε προβλήματα των δικτύων. Ε, χρειαζόμαστε ε, περισσότερα, δικ... περισσότερα ευφυή δίκτυα, διότι το δίκτυο στην Πορτογαλία μπορεί να φτάσει Καλύψει 100% των αναγκών μας, μπορεί να καλύψει 100% των αναγκών μας και τις ενέργειες που παράγεται από τις ανανεώσιμες ε, πηγές. Οπότε θέλουμε να πετύχουμε ε, ακριβώς αυτό το στόχο, το 15% που ανέφερε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τελευταία συμπεράσματά του, ε, για την διασύνδεση, την περισσότερη διασύνδεση και την αξιοποίηση των ευφυών δικτύων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Είπατε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Ιδίω εκεί μα είπατε για το ότι θέλετε η θέρμανση να μην ε, δημιουργεί του άνθρακο και στις και τις μεταφορές το ίδιο. Χθες μας κάλεσε το Ιώτα με έναν και άλλους συναδέλφους. Εδώ στις Βρυξέλλες. Είδαμε κάποια ευρυδικά αυτοκίνητα, κάποια ηλεκτρικά, κάποια ευρυδικά και σύντομα ελπίζουμε να έχουμε σε λογικές τιμές τέτοια αυτοκίνητα για όλο τον κόσμο. Έτσι όπως να τα εξηγήσατε και εσείς για τα ρητά καύσιμα, για τον αποκλεισμό τους από τις μεταφορές, για τα ανανεώσιμα τώρα. Ο συνάδελφος είπε για το θέμα της εύλογης τίμης. Για το διαλυπόμενο χαρακτήρα επίσης ακούσαμε. Και ξέρετε, στη χώρα μου ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για την αιωλική ενέργεια, τις σχετικές ε, τουρμπίνες. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Εγώ σε ευχαριστώ. Κύριε Βέρνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για αυτά τα οποία μας είπατε. Πράγματι στη Γερμανία έχουν φτάσει οι ανανεώσιμες πηγές θα έλεγα μία ισότητα τιμής, ίσως και κάτω εάν υπολογίσουμε το συνολικό κόστος της ανομικής ενέργειας. Και αν το υπολογίζαμε και αυτό θα αυξανόταν ακόμη περισσότερο το πραγματικό κόστος ατομικής. Ε, άκουσα να λέτε πως ε, χρειάζονται μια αποκεντρωμένη δομή δικτύου ε, οι ανανεώσιμες ενώ οι τωρινές τεχνολογίες σε ένα κεντρικό δίκτυο και έχουμε το πρόβλημα το ότι χρειαζόμαστε τις δύο αυτές δομές παράλληλα. Ποια μορφή λοιπόν θα μπορούσε να έχει η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές για να φύγουμε από τα παλαιά εργοστάσια ορυκτών πηγών ενέργειας και αυτό το οποίο είπε και ο συνάδελφος τις διασυνδέσεις γιατί οι ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα εάν έχουμε μία ενεργειακή ένωση και φτάσουμε αυτό το 50% των διασυνδέσεων. Σας ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Σας παρακαλώ κυρία μου. Παρατηρήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του εισηγητού και τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις ενδείξεις που μας δίνουν οι τιμές. Ό,τι αφορά τον άνθρακα. Η απάντηση είναι απλή. Οι τιμές EGS είναι σαν να δίνουμε στα παιδάκια σε ένα παιδικό πάρτι την ανταμοιβή του γιατί έπαιξαν καλά ένα παιχνίδι. Αλλά δεν επηρεάζει αυτό τις τιμές των ανανεώσιμων. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα στον EGS. Ε, Ούτε οι ανανεώσιμες χαίρονται γι' αυτό. Πρόσφατα ε, προσεκλήθην σε συναντήσεις με προσώπους ε, από την ε, βιομηχανία χάλιβα στην Ευρώπη και μου αρέσει να πηγαίνω τη μηχανή άνθρακα στην Ευρώπη, συγγνώμη, ε, και πηγαίνω σε αυτές τι συνεδριάσεις γιατί μου αρέσουν, αλλά βλέπουμε ότι τα ποσοστά χρήση χάλιβα και άνθρακα και αερίου δεν είναι εύκολο να αλλάξουν θα πρέπει να ε, δούμε αυτό που είπαν και άλλοι ομιλητές, όπως η κυρία Νίμπλερ, τις οποίες εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά στη Γερμανία. Εδώ θέλουμε εξυγχρονισμό ε, του συστήματος ενέργειας, κάτι που είναι η ραχοκοκαλιά για την υπόλοιπη κοινωνία μας και τη λειτουργία της. Ξέρετε ότι οι τιμές της ενέργειας είναι πολύ σημαντικές. Όχι μόνο για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στη Γερμανία, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Και έχουμε και ένα τέτοιο σύστημα στην ε, Γερμανία που εφόσον θέλουμε μια βιομηχανοποιημένη χώρα και το σύστημα της εντατικής χρήσης, αυτό είναι ένας κοινωνικός συμβασμός που γίνεται σεβαστός η τιμή για τον μεμονωμένο χρήστη μπορεί να διακυμαίνεται, αλλά ήδη τα περιθώρια της τιμής ε, μειώνονται, οπότε υπάρχουν σοβαρές διακυμάνσεις. Για τα συστήματα τώρα, και τις συνδέσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να τα επιλύσουμε όλα αλλά θα ήταν κρίμα, ε, διότι τα κράτη-μέλη ε, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαν να συνεργαστούν πολύ καλύτερα από ότι στο παρελθόν. Είναι λάθος μήνυμα να μην έχουμε δεσμευτικούς στόχους. Μπορούμε και πρέπει να έχουμε για την πρόσβαση στην αγορά. Ήδη στη Γερμανία Ο μηχανισμός ε, feed-in δεν χρησιμοποιείται κατά ένα 70%. Όμως ε, ε, και αυτό που είπαμε για το φαινόμενο των υποδομών, το login το λεγόμενο και εφόσον θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει παραδοσιακά. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια, αλλά όσο περισσότερες και ευφιέστερες πηγές, ανανεώσιμες πηγές έχουμε στο δίκτυο, τόσο καλύτερο θα είναι. Δεν είναι τίποτε δύσκολο. Δεν είναι τόσο μαγικό αυτό που σημαίνει στην εταιρεία μου. Ε, συνεργαζόμαστε με τις γερμανικές περιφέρειες και δήμους και κοινότητες. Εκεί ε, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά στην καθημερινότητα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι κάπω όμοιρα τη Γαλλία, αλλά οι δικέ μα οι περιοχές συνεργάζονται με γειτονικέ χώρε. Είναι απλό να ε, λειτουργήσει όμω αυτή η διασύνδεση αλλού. Ε, επίσης, πολλή έρευνα πρέπει να γίνει για να είναι ακόμη πιο ευφυές το δίκτυο στο μέλλον, να έχουμε συγκεκριμένε λύσεις και κυρίως στον εξοηλεκτρικό τομέα. Είναι πολλά αυτά που γίνονται, που τα έχουν ε, υλοποιήσει οι παλιοί μας ε, πάροχοι, ε, η ο φωτισμός σε συγκεκριμένους αυτοκινητοδρόμους. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτά. Και όταν λέτε στη χώρα μου έχετε μόνο 500 ώρες από την αιωλική, τι να σας πω, ε, είναι πολύ παλιά η τεχνολογία σας. Δεν μπορεί με έναν έξυπνο σχεδιασμό να έχετε τόσο χαμηλούς αριθμούς. Κάτι συμβαίνει στη χώρα σας. Στην ε, Γερμανία έχουμε σε συνεργασία με τη Δανία πάνω από 900 ώρες. Κάποιοι σας παραπληροφορούν και λυπάμαι που τα ακούω αυτά. Αυτό θα ήταν ένα μήνυμα που θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε πριν από 15 χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μπορούμε να τα δούμε και εκτός αν θέλετε. Αλλά οι ε, υποδομές. Το είπα ότι το πολύ καλό θα ήταν αν κοινοβούλιο ζητούσε από την Επιτροπή να ε, κάνει την ε, σωστή ανάλυση των αναγκών προς το αέριο. Διότι Νομίζω ότι έχουμε μια σειρά από κακές επενδύσεις, άχρηστες επενδύσεις. Δεν βοηθάμε έτσι ούτε τους μεγάλους παρόχους αερίου. Πρέπει να έχουν και αυτοί ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για να ασχοληθούν και με άλλες επενδύσεις, όπως με το ορυκτό πετρέλαιο. Και να πω ότι ο Πούτιν μας έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Το να κοιτάζουμε πώς θα του πάρουμε περισσότερο αέριο για να το φέρουμε εδώ είναι ξεπερασμένη προσέγγιση. Και για την υπερχρήση των ε, ανανεώσιμων. Όσο περισσότερε έχει ανανεώσιμε πηγέ κανεί στο δίκτυο, τόσο λιγότερο χρειάζεται το ε, πετρέλαιο και τα υπόλοιπα. Δεν είναι πρόβλημα να συνδυαστούν. Απλώς χρειαζόμαστε καλύτερες διασυνδέσεις και θιέστερο δίκτυο. Τα απαντήσατε όλα, λίγο πολύ, ναι. Ως προς το προσιτόν ε, των τιμών, νομίζω το κάλυψα. Ε, αν δείτε τη διαφάνεια από την παρουσίαση, τι ήδη πληρώνουμε στα offshore και στα inshore. Είχαμε μείωση τα τελευταία 15 χρόνια, χρόνο το χρόνο, στις ανανεώσιμες. Εάν λοιπόν ε, θέλουμε να ισχύει ένα 24ωρο, ε, θα έχουμε ακόμη λιγότερες πιέσεις, ακόμα λιγότερους περιορισμούς με τη μετακίνηση από αυτές τις υποδομές που έχουμε σήμερα προς κάτι άλλο. Νο, πραγματικά λοιπόν εκπλήσουμε κάποιες φορές και αν μπορώ να είμαι κάπως κοινική, εάν μου έδινε το management σε μια εταιρεία το έγγραφο που έχετε εσεί στα χέρια σα για να εργαστείτε με τέτοια επιχειρήματα, με τέτοια ε, ανάλυση, εγώ ω διεύθυνση τη εταιρεία μπορεί και να ζητούσα πτώχευση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κυρία μου για τι απαντήσει σα. Και σε ευχαριστούμε και για όσα μα είπατε και τώρα ήρθε η ώρα για την ε, σύνοψη, τη σύνθεση των όσων ε, συζητήσαμε. Ε, ακόμα έχουμε τους πέντε ομιλητές και τους ευχαριστούμε και πάλι. Άλλα θα δοθεί ο λόγος στον κύριο εισηγητή. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και να ευχαριστήσουμε όλους τους εκλεκτούμενους μας προσκεκλημένους ομιλητές. Νομίζω ότι δίνει η παρουσία τους όθηση στις εργασίες μας στην υπό σύνταξη έκθεσή μας μια που σήμερα με αυτές τις εισηγήσει και με τις ερωταπαντήσεις νομίζω ότι εφήξαμε όλα τα επιμέρους θέματα τα οποία καλύπτονται από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανέωσιμες ενέργειας, πυρηνική ενέργεια, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, βεβαίως δεν θα επισέλθω τώρα στις λεπτομέρειες. Σίγουρα η έκθεση θα καλύψει αυτές τις λεπτομέρειες και η συζήτησή μας θα συνεχιστεί. Και στην Επιτροπή και γενικότερα στο Κοινοβούλιο για όλα τα επιμέρους θέματα. Πάντως, σήμερα μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος. Οπότε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητάς για τις εισηγήσεις τους. Όμως έχω κάποιες γενικού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Όπως είπαμε στην αρχή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια αυθεντική στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη, δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να ε, αποσκοπεί στο να καλύψει τον επόμενο χειμώνα. Θα πρέπει να είναι κάτι πιο μακρόπνο. Και για μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα. Σήμερα προέκυψε ακριβώ ότι η ενέργεια είναι ένας τομέας όπου δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πολιτική επιρροή, επίδραση και τα, τις, τις, γεωπολιτικές μεταβλητές. Τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για την πυρηνική ενέργεια. Πάντοτε υπάρχουν πολιτικές εντάσεις που δημιουργούνται όταν ε, έχουμε να κάνουμε ενέργεια. Έτσι είναι η ζωή. Ναι. Οπότε καταρχήν δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το θέμα, άρα θα πρέπει να λάβουμε τις ορθές πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι θέμα του να αποπολιτικοποιήσουμε τη στρατηγική, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να λάβουμε υπόψη τις τεχνικές πτυχές, την οικονομική ανάλυση, τις πολιτικές θέσεις, τους πολιτικούς στόχους. Εν κατακλείδη, σαν συμπεράσματα, σαν μάθημα από τη σημερινή συζήτηση, ας ε, λάβουμε υπόψη το εξής. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα της στρατηγικής για, για ενεργειακή ασφάλεια. Θέλουμε να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εξαγωγές. Όμως τα προγνωστικά λένε ότι θα αυξηθεί η εξάρτηση. Εμείς όμως θέλουμε να την μειώσουμε. Άρα θα συνεχίσουμε να είμαστε εξερτημένοι. Ασφάλεια τι είναι επομένως το να γίνει κατανομή του βάρους της εξάρτησης. Κάθε αυτή η εξάρτηση δεν είναι πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση, μια διασπορά αυτής της εξάρτησης. Να μην έχουμε μόνο μια πηγή οπότε να έχουμε μονόπλευρη πολιτική επιρροή στην Ευρώπη. Να, τι πάει να πει, αλληλεγγύη. Υποδομές, αγορές, δυνατότητα κατανομής αυτού του βάρους για τα κράτη-μέλη, κατανομή του βάρους από οτιδήποτε πρόκειται από το εξωτερικό σαν βάρος. Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους όσους μας ομίλησαν. Μεγάλη βοήθεια ήταν αυτό για τη δουλειά μας. Θα συνεχιστεί η προβληματική και η συζήτηση. Ο Πρόεδρος, όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα τρίγωνο ενεργειακό. Ξεκινήσαμε από την ασφάλεια. Θεωρούμε ότι η περισσότερη ασφάλεια σημαίνει περισσότερες δυνατότητες για χαμηλές τιμές ενέργειας, ανταγωνιστικές τιμές. Ίσως αυτό δεν είναι καλά μαντάτα για τις ε, εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην ε, ενέργεια. Τον ένα δηλαδή χαμηλότερες τιμές, αλλά είναι καλά μαντάτα για τις ΜΜΕ, για τους πολίτες, για τη στρατηγική έξοδο από την κρίση, και, αλλά και για το περιβάλλον προφανώς. Πρόκειται μόνο για την αρχή της διαδρομής. Στις 3.12 θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα συζητήσουμε τα της έκθεσής μας για την ε, στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια. Ανταλλαγή απόψεων. Σε ένα μήνα. Σα ευχαριστώ. Αλλά πρώτα πρώτα οι εισηγητές μας. Δύο βρίσκονται εδώ ακόμη στο Προεδρείο κ. Σέλνας κ. Φουκέ και έχουμε τρεις άλλους. Τον καθηγητή κ. Μπάρτη, τον κ. Μπαρτούσκα και τον κ. Σπέντας εδώ βρίσκονται ακόμη μεταξύ μας. Οπότε όλους τους ευχαριστούμε για τη συζήτηση, για τα όσα είπαν και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον για να ξαναανταλλάξουμε απόψεις. Και πάλι ευχαριστούμε. And, uh, next part of our meeting. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση στις 3 η ώρα μετά το σύντομο διάλειμμα. Ευχαριστώ.